Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε. Ας αρχίσουμε με το πρώτο σημείο της μέσας διάταξης, δηλαδή την έγκριση της μέσας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, ας εγκρίνουμε χωρίς τροποποίηση τη μέσα διάταξη. Δεύτερο σημείο είναι η έγκριση των πρακτικών από τη συνεδρίαση της 14ης Δεκεμβρίου 16-17 Μαρτίου. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις με τα τέλη της συνεδρίασης, θα εγκριθούν τα πρακτικά. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Αρχικά για την αποστολή στην Ιρλανδία. Τα πρακτικά της αποστολής Μπορείτε να τα βρείτε και στο φάκελο της ε, συνεδρίασης. Έχουμε διερμηνία σε 21 γλώσσες και ως ε, ήθιστε <coughs> και ο φάκελος ε, διατίθεται και ηλεκτρονικά στην εφαρμογή e-meeting και η συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω διαδικτύου. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο τέταρτο σημείο, ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Καρμένου Βέλλα, Επίτροπο Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλίας, ως ε, τμήμα του ε, διαθετημένου διαλόγου. Αρχικά θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω και να σας υποδεχθώ εδώ. Καλώς ήρθατε κύριε Βέλλα στη σημερινή συνεδρίαση. Όπως ξέρετε αυτή η συνάντηση λαμβάνει μέρος στο πλαίσιο του διαλόγου μας με την Επιτροπή. Σε αυτό το πλαίσιο Θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια σε ό,τι φορά την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας για το 2016 και της ε, προτεραιότητά σας ε, πέραν του 2016. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι περισσότερο για τις προτάσεις σας ε, σε ό,τι αφορά την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, το θεματολόγιο 2030 για την i4 ανάπτυξη και το συνεχιζόμενο έλεγχο fitness check. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα ήθελαν επίσης να ακούσουν ε, κάτι για το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της ε, ελαφροθυρίας, ε, κατά της διάβρωσης των δασών και συνεχιζόμενων νομοθετικών φακέλων σε ό,τι αφορά τις εκπομπές του άνθρακα και άλλα τέτοια ζητήματα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Έχετε το λόγο για τα εισαγωγικά σας σχόλια και μετά θα γίνει και συζήτηση με τους συναδέλφους μας. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ Τζοβάνι. Καλό απόγευμα σε όλους τους ευρωβουλευτές και συναδέρφους και όπως είπατε θα ήθελα να περάσω κατευθείαν στα βασικά σημεία του προγράμματός μας. Οτιδήποτε ξεχάσω ε, μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Μπορεί να θυμάστε ότι στην ακρόασή μου εδώ στο Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2014 είπα ότι το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον ε, θα είναι το πλαίσιο προσανατολισμού μου. Το 7ο αυτό πρόγραμμα ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Παρακολουθώ στενά τις εργασίες και χαίρομαι που μπορώ να πω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ καλό όσον αφορά τις, ε, ε, τους εννέα στόχους προτεραιότητας του προγράμματος και Έχω εξαιρετικές ε, εργασιακές σχέσεις ε, και με πολλούς ε, από εσά προσωπικά, αλλά και με το σύνολο του Κοινοβουλίου πάνω σε πολλά θέματα. Το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στις 10 προτεραιότητες του Προέδρου Γιούνκερ και επικεντρώνομαι κυρίω σε τρει τομεί. Πρώτον, ε, πράσινο προσανατολισμό, οικολογικό προσανατολισμό τη Οικονομία, Δεύτερον, ε, καλύτερη επαφή με του πολίτε. Και τρίτον, να αναλάβουμε δράση, making it happen. Θα αναφερθώ σε αυτού του τρει τομεί ε, κατά σειρά, αλλά θα ήθελα πρώτα να αναφερθώ σε δύο σημαντικέ εξελίξει στο δεύτερο εξάμεινο του 2015. Αναφέρομαι στο θεματολόγιο αηφόρου ανάπτυξης 2030, μαζί με την Διεθνή Συμφωνία για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής ε, στο COP21 στο Παρίσι, που αποτελούν ε, δύο ε, ορόσημα στην παγκόσμια προσπάθεια για καλύτερη αηφορία. Όσον αφορά το θεματολόγιο 2030, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επίτευξη τόσο φιλόδοξου αποτελέσματο στι ε, διαπραγματεύσει ε, για το θεματολόγιο 2030 και θα συνεχίσουμε ε, αποφασιστικά να παίζουμε ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή και παρακολούθηση τη εφαρμογή των 17 στόχων αηφόρου ανάπτυξης και τους 169 επιμέρους στόχους. Όπως γνωρίζετε, προβλέπουμε το 2016 μια πρωτοβουλία για τα επόμενα βήματα όσον αφορά το ευρωπαϊκό μέλλον ε, που θα συνδέει την εφαρμογή των ε, στόχων αηφορίας ε, με την αναθεώρηση Ευρώπη 2020 για να έχουμε οικονομική ανάπτυξη καθώς και κοινωνική και περιβαλλοντική αηφορία. Θα εργαστούμε σε δύο φάσεις εντός του έτους θα εκδώσουμε ανακοίνωση που χαρτογραφεί τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές για την ε, εφαρμογή των στόχων αηφορίας, ε, καθώς ε, και τις σχετικές πρωτοβουλίες, όπως είναι η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινή Αντίληψης για την Ανάπτυξη ή της δουλεια της Eurostat για την παρακολούθηση της αηφόρου ανάπτυξης. Με βάση αυτές τις εργασίες θα ασχοληθούμε με μια στρατηγική για την Ευρώπη μετά το 2020. Θέλουμε η διαδικασία αυτή να είναι όσο γίνεται πιο συμμετοχική και να κινητοποιήσουμε όχι μόνο τους εμπειρογνώμονε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αλλά να υποφεληθούμε και από τις δικές σας εμπειρίες, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων. οι πρώτες ε, κατευθυντήρες γραμμές ε, για τα θέματα αυτά θα συζητηθούν από το Σώμα των Επιτρόπων φέτος τον Ιούλιο όσον αφορά την, ε, την πράσινη ανάπτυξη. Θέλουμε να διασφαλίσουμε οι οικονομικές μας δραστηριότητες ε, να είναι βιώσιμες, ε, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση όχι μόνο για να πετύχουμε τους στόχους για την αηφόρο ανάπτυξη, αλλά θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει και κάποιες πιο μακροπρόθεσμες προκλήσεις. Η Ευρώπη δεν έχει πολλούς φυσικούς πόρους, έχει όμως ε, γνώση και δεξιότητες. Θέλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε την αξία εντός της οικονομίας όσο γίνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αυτό η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να εντείνουμε την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης εντός της Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη είναι επικεφαλής ε, στον τομέα αυτών, ε, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ε, τα τελευταία στοιχεία μας δείχνουν ότι έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα ως προς τους πόρους την τελευταία δεκαετία και βλέπουμε να υπάρχουν τάσεις για μια πιο αηφόρο κατεύθυνση, αλλά απομένουν πολλά να γίνουν ακόμα για να αποσυνδέσουμε τα θέματα των πόρων από την οικονομική ανάπτυξη. Η πράσινη ανάπτυξη στο πλαίσιο της ε, στρατηγικής Ευρώπη 2020 σημαίνει μείωση του κόστους ε, των υλικών ε, και την μείωση της ζημιάς στο περιβάλλον, ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Μιλάμε δηλαδή για την κυκλική οικονομία. Πέρσι τον Δεκέμβριο παρουσιάσαμε πολύ καλά αποτελέσματα υιοθετώντα μια νέα στρατηγική για κυκλική οικονομία. Εάν εφαρμοστεί πλήρω η στρατηγική αυτή, θα έχουμε τριπλό κέρδο για την κοινωνία, θα έχουμε εξοικονόμηση για τι επιχειρήσει Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργία θέσεων απασχόληση και μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων ε, συμπεριλαμβανομένων των ε, ανθρακούχων εκπομπών. Τώρα επικεντρωνόμαστε κυρίω ε, στα διάφορα στοιχεία που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων. Επίσης, ε, έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του σχεδίου δράσης ε, πέρσι. Ε, ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του Horizon 2020, βιομηχανία 2020 στην κυκλική οικονομία και η Κομισιόν υιοθέτησε την πρότασή τη για την επιγραμμική πώληση αγαθών και πριν ένα μήνα, ακριβώς στι 17 Μαρτίου, παρουσιάσαμε έναν αναθεωρημένο κανονισμό για τα λοιπάσματα που συμπεριλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά για βιολογικά ε, λοιπάσματα και λοιπάσματα που βασίζονται σε βιοαπόβλητα. Τώρα ε, ετοιμάζουμε ένα νέο πρόγραμμα δράσης οικολογικού σχεδιασμού. Εξετάζουμε δηλαδή την ενεργειακή απόδοση των ε, προϊόντων, ε, αλλά ε, επίσης σε τι βαθμό είναι δυνατόν να επισκευαστούν, να ανακυκλωθούν και να αναβαθμιστούν. Επίσης, η δέσμη μέτρων προβλέπει έκθεση πρόοδου πέντε χρόνια μετά την υιοθέτησή της. Ωστόσο, συζητάτε να γίνονται πιο συχνές επικαιροποιήσει ε, και ενημέρωση των κρατών μελών ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων ενδιαφερομένων. Οι συζητήσεις για τις ε, νομοθετικές προτάσεις για τα απόβλητα έχουν ξεκινήσει πολύ θετικά και για τη δράση στα κράτη-μέλη και στο, στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου ήταν θετική. Προσλέπω στην ε, συνεργασία μαζί σας, ξεκινώντας από την ε, παρουσίαση της έκθεσης από την εισηγήτρια την Σιμώνα Μποναφέ τον Μάιο στην Επιτροπή σας ε, και την υιοθέτηση τον Νοέμβριο. Ήδη έχουν γίνει κάποιες προπαρασκευαστικές συναντήσεις με την Σιμώνα και το προσωπικό της, καθώς και με τους σκιώδεις εισηγητές. Προσφέρουμε την πλήρη συνεργασία μας και τις τεχνικές συμβουλές μας για τους επόμενους μήνες. Επίσης, τα θαλάσσια απόβλητα είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Πρέπει να ε, βρούμε μια προσέγγιση ώστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και στη στεριά και στη θάλασσα. Ήδη υπάρχουν καλές πρωτοβουλίες, ε, καθαρισμός ε, ακτών, αλληλεία απορριμμάτων και θα πρέπει να μειώσουμε την χρήση των πλαστικών σακουλών μιας χρήσης αλλά πρέπει να είναι πιο καλά ε, συντονισμένες αυτές οι δράσεις. Ε, οι, ε, τα απορρίμματα, τα απόβλητα είναι μόνο ένα μέρος του κύκλου. Χρειάζονται λοιπόν στοχευμένες επενδύσεις στον τομέα αυτών. Θα ήθελα να αναφέρω ότι η πράσινη εβδομάδα της φετινής χρονιάς τέλη του Μαΐου θα είναι αφιερωμένη στις επενδύσεις για ένα πιο πράσινο μέλλον θα πρέπει να φροντίσουμε το οικονομικό μας σύστημα να προωθεί την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και να μας βοηθήσει να πετύχουμε τις ε, δεσμεύσεις που κάναμε πέρσι στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη για το θεματολόγιο 2030, καθώς ε, και στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο συμμετέχει προορατικά στο πρόγραμμα της Πράσινης Εβδομάδας και θα χαρώ πολύ να δω όσο γίνεται περισσότερος από σας εκεί. Όσον αφορά το φυσικό κεφάλαιο, η βιοπικιλότητα αποτελεί πόρο από μόνο παρότι δεν είναι πάντα πολύ ορατή. Το φυσικό κεφάλαιο και τα οικοσυστήματα μας παρέχουν καθαρό νερό, ε, ε, επικονίαση των φυτών, ε, γεωργική παραγωγή και αποτελεί στήριγμα για την οικονομία μας, την κοινωνία μας και αποτελεί προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ευημερία μας. Εάν λοιπόν ε, δεν φροντίσουμε τα οικοσυστήματά μας, θα χάσουμε αυτούς τους πόρους και ε, απαιτείται πολύ χρήμα και πολύς χρόνος για να αντικαταστήσουμε ε, με τεχνητές λύσεις. Έτσι λοιπόν η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί δαπάνη, αποτελεί εξοικονόμηση και επένδυση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον η ενδιάμεση αναθεώρηση της ε, Κομισιόν, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και η έκθεση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, όλα στέλνουν ένα σαφές μήνυμα όσον αφορά την μεγάλη σημασία ενίσχυσης των προσπαθειών μας για να πετύχουμε τους στόχους βιοποικιλότητας για το 2020. Τέσσερα χρόνια όμως πριν από την ημερομηνία αυτή δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε το στόχο μας. Ε, θα είναι απαραίτητο να έχουμε περισσότερη πολιτική συνοχή και τομεί όπω είναι η γεωργία και η δασοκομεία που μαζί καλύπτουν το 80% των εδαφών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βρίσκονται στον πυρήνα της λύσης για να αναχαιτήσουμε την απώλεια βιοπικιλότητας. Λέγεται μερικές φορές ότι κάτι που δεν μπορεί να μετρήσει κανείς δεν θα συμβεί. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε πιο ορατή την αξία της φύσης, να γίνει πιο κατανοητή και να ενσωματώσουμε τη διάσταση αυτή στη λήψη αποφάσεων και στον προγραμματισμό μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό βήμα για να αντιμετωπίσουμε έναν, μια από τις βασικές αιτίες απώλειας της βιοπικιλότητας ήταν η, η, η υιοθέτηση του κανονισμού ε, για τα... Ε, τα χωροκατακτητικά είδη. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσά πιστεύουν ότι βιαστήκαμε πολύ. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες ώστε να μπορέσουμε να επικαιροποιήσουμε τον κατάλογο των ειδών αυτών ε, εντός της χρονιάς. Σε ό,τι αφορά το fitness check για τη ε, φύση, στα, στη συνέχεια της χρονιάς θα παρουσιάσουμε και ε, την συνέχεια σε ό,τι αφορά το fitness check της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας προ τη φύση. Ε, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και σε ό,τι αφορά τους πολίτες αλλά και τα ενδιαφέροντα μέρη. Η διαβούλευση έλαβε περισσότερες ε, απαντήσεις από ό,τι εκείνη για το TTIP και αυτό δείχνει ότι η φύση πραγματικά είναι ένα σημείο μεγάλου ενδιαφέροντο για τους πολίτες. Η απόφαση διεξαγωγή ενό ε, fitness check για τι δύο οδηγίε για τη φύση Αναγνωρίζω ότι αυτέ οι δύο νομοθετικέ πράξει ε, έχουν τεθεί σε ισχύ εδώ και πολλά χρόνια και έχει έρθει η ώρα να ελέγξουμε κατά πόσο λειτουργούν σωστά και αν μπορούν να βελτιωθούν. Ε, Αυτό ο έλεγχο το fitness check, θα μα βοηθήσει να κατανοήσουμε τι πηγαίνει καλά, τι όχι και γιατί. Βρισκόμαστε τώρα στα τελευταία στάδια του fitness check και θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα σε μια συνδιάσκεψη για τη φύση στην Ευρώπη, η οποία διοργανώνεται από τις κάτω χώρες στα τέλη της Προεδρίας της. Στη συνέχεια του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προτείνει συγκεκριμένε δράσει ε, για την συνέχιση του fitness check, όπω έχουμε ορίσει και στο πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2016. Σήμερα, δυστυχώ, ε, δεν μπορώ να ανακοινώσω τα αποτελέσματα τη Επιτροπή ό,τι αφορά το fitness check, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το εγχείρημα. Όμω, θέλω να είμαι σαφή, δεν ε, προτίθεμαι να προτείνουν οποιαδήποτε μείωση και υποβάθμιση των στόχων ε, της νομοθεσία που ε, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής. Όπως ανέφερε και ο Τζοβάνι, ε, θα θέλατε να ακούσετε κάτι και για το παράνομο, εμπορία ε, άγριων ζώων. Εργαζόμαστε για την διατήρηση ειδών και οικοσυστημάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παγκοσμίω όμω βλέπουμε μια δραματική αύξηση τη ελευθερία. Βλέπουμε ότι μόνο 20.000 ε, ελέφ... μάλλον ε, το 2013 μόνο, πάνω από 20.000 ε, ελέφαντες έπεσαν θύματα αυτού του παράνομου κυνηγιού. Και αυτό δεν καταστρέφει μόνο ζωές και θέτει σε κίνδυνο τα ήδη επαπειλούμενα είδη, όμως ε, και χρηματοδοτεί το έγκλημα ε, και στερεί από τις τοπικές κοινότητες, τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, ένα πολύ σημαντικό εισόδημα. Αλλά είναι και η ανθρώπινη τραγωδία με στη μέση, γιατί και πολλοί άνθρωποι κάνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να προστατεύσουν αυτά τα είδη. Η Επιτροπή απάντησε στις 26 Φεβρουαρίου με ένα ολοκληρωμένο και εύρωστο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της, του φαινομένου αυτού. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό και έτσι υπάρχει σαφή ανταπόκριση και προς ε, την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ώστε η Ευρώπη να κάνει κάτι για αυτό το ζήτημα. Οι πρώτε ε, αντιδράσει των κρατών μελών είναι θετικέ και αναμένουμε ότι το Συμβούλιο Περιβάλλοντο θα υιοθετήσει το σχέδιο δράση στην συνάντηση του Ιουνίου και περιμένω με ενδιαφέρον και την έκθεση της Επιτροπής σας για αυτό το ζήτημα. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει ε, ένα σημαντικό αριθμό δεσμεύσεων που είναι όλοι <laughs> σημαντικές και είναι σημαντικό να υλοποιηθούν εντός του χρονοδιογράμματος, ούτως ώστε να υπάρξει ε, απτή πρόοδος. Έχουμε αρχίσει την υλοποίηση του προγράμματος και ε, θα συζητήσουμε περαιτέρω με τα κράτη-μέλη πώς μπορούμε να περαιτέρω να προωθήσουμε την υλοποίησή του. Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η συνδιάσκεψη των μερών της Σύμβασης ε, για το Διεθνές Εμπόριο των ε, Επαπειλούμενων Ειδών. Η Σύμβαση ΣΥΤΕΣ το Σεπτέμβριο και βασιζόμαστε και στη δική σας στήριξη που είναι κρίσιμη σημασία ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να τεθεί επικεφαλής των προσπαθειών για την εξάλληψη του φαινομένου ε, αυτού σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη σύνδεση με τους πολίτες. Οι υπερβαλλοντικέ πολιτικές αποτελούν απόσπαστο τμήμα για την διασφάλιση της μια αηφόρου οικονομίας μακροπροθέσμώ, όμως είναι σημαντικέ και για του πολίτε μας, γιατί ε, άπτονται πολλών πλευρών τη καθημερινότητάς τους. Στην ακρόασή μου ενώπιόν σας για να λάβω ε, το χρήσμα του Επιτρόπου και εγώ σας ανέφερα πολύ συγκεκριμένα τις προτεραιότητές μου ε, για την διασφάλιση ε, και των ζωών και της υγείας ε, των ε, πολιτών μας και την προστασία μας απέναντι στους, ε, στους κινδύνους για την υγεία. Και η περιβαλλοντική πολιτική λοιπόν είναι πολύ σημαντική για αυτό το σκοπό. Σήμερα πάρα από το 99% του πόσιμου νερού που τροφοδοτείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασφαλές χάρη στη συνεχή βελτίωση της υλοποίησης ε, τη Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Δυστυχώ δεν μπορούμε να πούμε και το ίδιο για την ποιότητα της ατμόσφαιρας που αναπνέουμε στην Ευρώπη. Ε, η δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την καθαρή ατμόσφαιρα έχει ως στόχο να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των πρόωρων θανάτων που οφείλονται στην ε, ατμοσφαιρική ρήπανση στην Ευρώπη και να περιορίσει σημαντικά τις ασθένειες του αναπνευστικού, ενώ παράλληλα θα εξοικονομήσει έως και 140 δις ευρώ σε δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης έως το 2030. Εκτιμώ τις πολύ σημαντικές προσπάθειες της συναδέλφου μας ε, Julie Gerling και των σχεδόν ε, εισηγητών ε, για να καταλήξουμε σε μία συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για την οδηγία για, τις, για τα εθνικά όρια εκπομπών. Εάν καταφέρουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, μπορούμε να καταδείξουμε πόσο σημαντική είναι και η ευρωπαϊκή πολιτική για τα, σε ό,τι αφορά τα ωφέλη στην υγεία των ευρωπαϊκών πολιτών. Αλλά και σε ό,τι αφορά την ε, σύμβαση ε, Μιναμάτα για το ψευδάργυρο έχουμε πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά ωφέλη αλλά και στον τομέα της υγείας γιατί έτσι έχουμε ε, μειωμένη έκθεση σε ψευδάργυρο παγκοσμίω αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να ε, θέσουμε τέλος ε, στην ε, παρασκευή προϊόντων με χρήση και εμπορία ε, ψευδαργύρου και να απαγορεύσουμε οποιαδήποτε χρήση ψευδαργύρου στους, σε προϊόντα και στη βιομηχανία εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτό και αν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία τη υγεία και του περιβάλλοντο. Τα όσα η Κομισιόν πρότεινε στι αρχέ ε, του Φεβρουαρίου σημαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ηγείται τη παγκοσμία πολιτική υδραργύρου. Και είναι σημαντικό να κυρώσουμε την σύμβαση πριν τη θέση σε ισχύ ε, το αργότερο στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Αυτό απαιτεί ταχύτατε εργασίες από τους νομοθέτες και είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα. Πέραν του υδραργύρου, οι πολίτες προβληματίζονται σε ό,τι αφορά τις χημικές ουσίες ε, σε σύνδεση με πιθανό αντίκτυπο στην υγεία τους και στο περιβάλλον η αναθεώρηση REACH το 2017 αλλά και το fitness check όλη τη νομοθεσία που άπτεται των χημικών ουσιών θα ε, μας δώσει πολλά στοιχεία για την στρατηγική που θα εκπονηθεί το 2018 για ένα μη τοξικό περιβάλλον ε, το οποίο εντάσσεται και στο 7ο EAP. Ε, θέλω να καταδείξω ότι το επίκεντρο στην απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη δεν έρχεται σε αντίθεση με την περιβαλλοντική προστασία των σημερινών και μελλοντικών γενεών Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει όλα αυτά να πηγαίνουν ε, μαζί. Τώρα, πώς θα γίνουν όλα αυτά. Όλα αυτά τα ωφέλη και η αηφόρος ανάπτυξη, η βελτιωμένη υγεία και ευημερία και ε, ο περιορισμό των κινδύνων μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν οι πολιτικές και η νομοθεσία που ε, υιοθετούμε και εγκρίνουμε υλοποιούνται στην πράξη και σωστά. Και έτσι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το χάσμα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση στην Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και τρίτες χώρες ε, θα αναλάβουν φιλόδοξες πρωτοβουλίες. Πρέπει να έχουμε όμως και τα κατάλληλα εργαλεία, τα οποία να είναι επίκαιρα και κατάλληλα προς αυτό το σκοπό. Ε, και όλα αυτά τα παίρνουμε πολύ σοβαρά. Ήδη έχουμε διεξακάγει αξιολογήσεις ε, διαφόρων νομοθετικών πράξεων στον τομέα του περιβάλλοντος. Και θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Έχω ήδη αναφέρει το fitness check για τη φύση. Μια άλλη σημαντική αξιολόγηση που εκπονείται αυτή τη στιγμή έχει πιο εγκάριστο χαρακτήρα και συνδέεται με την, με την υποβολή περιβαλλοντικών εκθέσεων. Στόχος είναι οι εκθέσεις να είναι πιο σαφείς, επίκαιρες και εύκολες στην προετοιμασία τους. Και αυτό θα μεταφραστεί σε καλύτερα αποτελέσματα στην πράξη και χαμηλότερο διοικητικό άκθος για τις επιχειρήσεις. Η διαβούλευση ενδιαφερμένων μερών που κάναμε έχει ήδη οδηγήσει σε πολλές θετικές ιδέες και θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα το 2017 είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβλέπει την ε, σωστή υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας και δεν θα διστάσουμε να αξιοποιήσουμε και τις ε, ε, εξουσίες υλοποίησης της νομοθεσίας που μας εκχωρούνται από τις συνθήκες και να κινήσουμε διαδικασίες επιπαραβάση, παραβάση, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Βεβαίως, καλό θα ήταν να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Μία συμπληρωματική λύση είναι να καταγράφουμε την πρόοδο ε, και να προσπαθούμε να επιλύουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση υφιστάμενων αλλά και νέων δεσμεύσεων. Γι' αυτό και αναπτύσσουμε ε, το λεγόμενο EIR, ε, την αναθεώρηση της υλοποίησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που θα δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα σε ό,τι αφορά ε, την υλοποίηση ε, της νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη, κατά προτίμηση πριν τεθούμε σε διαδικασία επιπαραβάση. Θέλουμε να βελτιώσουμε ε, τη γνώση μας ό,τι αφορά τα εφιστάμενα κενά στην εφαρμογή της νομοθεσίας σε κάθε κράτος μέλος. Θέλουμε να δώσουμε νέες λύσεις και επιπροσθέτως αλλά και συμπληρωματικά προς ε, την ε, υλοποίηση του νόμου και εφαρμογή του νόμου. Θέλουμε να επισημάνουμε ε, τις κύριες αιτίε αυτών των χασμάτων, των κενών και να δώσουμε κίνητρα για την ανταλλαγή των πρακτικών. Ως πρώτο βήμα θα έχουμε εκθέσεις αναχώρα που θα προετοιμάζουν τον ε, τον διμερή διάλογο μεταξύ Κομισιών και κράτους μέλους. Αυτό θα επιτρέψει συζητήσεις ψηλού επίπεδου σε οποιαδήποτε σημαντικά τέτοια κενά που είναι και κοινά σε επιμέρους κράτη-μέλη. Δεν είναι μια νέα ιδέα αυτή έχουν υπάρξει αντίστοιχες ε, επισκοπήσεις στο παρελθόν σε άλλους τομείς πολιτικής, όπως είναι η νέα αγορά, η ψηφιακή οικονομία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χορολόγηση, προστασία του καταναλωτή και είχαμε μεγάλες επιτυχίες σε όλους αυτούς τους τομείς. Πριν τα τέλη του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στόχο ε, να παρουσιάσει και μια πρωτοβουλία για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Έτσι θα έχουμε ερημερευτικής κατευθυντήριες γραμμές σε ό,τι αφορά τις ε, αποφάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές θα βοηθούν τα κρατημέλη, τα εθνικά δικαστήρια και τους πολίτες, καθώς και περιβαλλοντικές ΜΚΟ, για να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις νόμιμες προκλήσεις. Για τις διεθνείς σχέσεις, δεν μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερο περιβάλλον στην Ευρώπη μέσω μόνης της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει τα κράτη να αναλάβουν δράση, να προχωρήσουν προς πιο κυκλικά οικονομικά πρότυπα, να υιοθετήσουν ατμοσφαιρικά πρότυπα εκπομπών, να καταπολεμήσουμε την εμπορία ανθρώπων, να ενισχύσουμε την ε, διαφορετικότητα και την βιοπικιλότητα και να περιορίσουμε τους ρήπους. Πρέπει να αυξήσουμε τη συνεργασία μας με ε, εταίρους κλειδιά και διεθνείς οργανισμούς και φέτος ε, θα έχουμε δύο σημαντικές ευκαιρίες να το κάνουμε αυτό. Έχουμε την συνεδρίαση των ε, μερών της Σύμβασης Βιοπικιλότητας και Απειλουμένων Ειδών αλλά θα πρέπει να ενισχύσουμε ενεργά την αποτελεσματικότητα στην κυκλή οικονομία μέσω του G7 και της, ε, του περιφερειακού outreach, των διμερών μάλλον outreach. Έχουμε επίσης την ανακοίνωση ακτικής πολιτικής, ε, μία λέξη θα πω. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι η παριθμόν ένα προτεραιότητα των ε, ενεργών πολιτικών της Κομισιόν και η επερχόμενη ανακοίνωση Κομισιόν για την Αρκτική θα τονίσει την βιώσιμη ανάπτυξη που θα πρέπει να εφαρμόσουμε στην περιοχή, το οποίο θα πρέπει να μεταφραστεί σε απτές δράσεις. Εγώ υπολογίζω στην ε, ενεργό συμμετοχή και στήριξή σας. Και για να ολοκληρώσω, προσβλέπω στην συνεχιζόμενη συνεργασία μαζί σας. Το στρατηγικό πλαίσιο είναι σαφές και τώρα πρέπει να περάσουμε από το σχεδιασμό και να περάσουμε στην υλοποίηση και στην εφαρμογή των δράσεων αυτών και διεθνώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενσωματώσουμε τις SDGs στις εσωτερικές και εξωτερικές μας πολιτικές, να εφαρμόσουμε τον κύκλο, την, ε, το, τη δέσμη κυκλικής ε, οικονομίας και να εφαρμόσουμε τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Όπως θέλουμε και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να ζουν σε ένα υγιή πλανήτη με υγιή τρόφιμα και νερό, με προϊόντα τα οποία θα έχουν προστατευτεί και θα είναι ασφαλές να τα χρησιμοποιήσει κανείς και σε ένα κόσμο με ένα ποικίλο οικοσύστημα στο οποίο δεν θα σπαταλούμε πόρους. Νομίζω ότι μπορούμε εντός των ορίων που μας θέτει ο πλανήτης μας να ζήσουμε αρκετά καλά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να ξεκινήσουμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ο Καρλ Χάινς από το ΕΛΚ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που τηρήσατε τον πρώτο κανόνα Κατά την ακρόασή σας εδώ υποσχεθήκατε ότι ε, θα έρχεστε τακτικά και πράγματι το κάνετε αυτό και θα ήθελα να σας επενέσω γι' αυτό. Ε, μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Προσπάθησα να ακούσω με προσοχή αυτά που είπατε. Και σκέφτηκα ότι α, ωραία, ε, βγαίνει ο ήλιος ε, όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα πάνε καλά τώρα. Έχω χτυπήσει πολλές φορές ε, στον τοίχο στις Βρυξέλλες ε, και δεν πιστεύω πια τα πάντα, αλλά πιστεύω αυτά που είπατε όσον αφορά τον έλεγχο καταλληλότητας στο fitness check κλπ. Εάν όμως ε, δούμε τι κάνει ο οργανισμός για το περιβάλλον τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές χώρες, μεταξύ άλλων και η δική μου μάλλον, που δεν ξεκινούν καν να εφαρμόζουν ε, τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δεν ασκηθεί απ' έξω πίεση σε αυτές τις χώρες, ε, δεν θα πετύχουμε αποτελέσματα. Και Έχω πει πολλές φορές ε, δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε πολύ μακριά. Ε, ας κοιτάξουμε τι γίνεται στις γειτονικές μας χώρες. Ε, στη δική μου χώρα έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τα λοιπάσματα. Νομίζω λοιπόν κύριε Επίτροπε ότι θα πρέπει να αναρωτηθείτε τι γίνεται όσον αφορά την ε, οδηγία που λέει ότι μέχρι το 2020 θα πρέπει να ανακυκλώνεται το 50% των απορριμμάτων. Ε, είναι κακή η κατάσταση και επιπλέον ε, δεν είναι πολύ σαφές τι εννοούμε όταν μιλάμε για ανακύκλωση. Άλλος το εξηγεί με τον ένα τρόπο, άλλος το εξηγεί με τον άλλον τρόπο. Χρειάζεται Λοιπόν, μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να κοινοτυπήσουμε τις κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν το ελάχιστο. Μία τελευταία παρατήρηση. Έχουμε τέσσερις εκθέσεις για την πολιτική απορριμμάτων. Ε, δεν έχω πολλά να επικρίνω εκεί, αλλά ε, εκπονήθηκαν οι εκθέσεις αυτές διότι δεν έχει ασκηθεί σωστά η πολιτική. Δεν έχουμε σωστή πολιτική για τη ε, διάθεση των απορριμμάτων στην Ευρώπη. Η μεγάλη μου επιθυμία λοιπόν είναι να ε, ασκηθεί περισσότερη πίεση Ευχαριστώ τον Επίτροπο για την εξαιρετική παρουσίασή του, τον ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ, τον ευχαριστώ για την καλή του βούληση, αλλά χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλους 50 ανθρώπους. Ε, ο προκάτοχός σας μου το είπε αυτό. Χρειαζόμαστε 50 ανθρώπους παραπάνω για να ελέγχουν την κατάσταση και η ε, κακή εδώ δεν είναι ο Γιούνκερ, είναι τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να ελεγχθούν. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πότση για την Σοσιαλιστική Ομάδα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο που είναι μαζί μας για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων και τη συζήτηση που είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Ε, χαίρομαι που αναφέρατε την ε, στρατηγική σε 2020 και είχαμε αποτύχει στον πρώτο έλεγχο του 2010. Δεν θέλω να επαναλάβουμε αυτή τη δυσαρεστή εμπειρία. Έχουμε ακόμα τέσσερα έτη εγώ δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξο για τα παραδοτέα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε την άποψή σα για δύο-τρία πράγματα. Αναφέρατε τα χαρακτηριστικά ήδη. Έχουμε <clears throat> νομοθεσία, αλλά η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως και αποτελεσματικά. <clears throat> Μπορούμε να παριθμίσουμε αντιρρήσεις και υπάρχουν επιχειρήματα και τα αναφέρατε, αλλά παραμένει μια ερώτηση. Εμείς τιμούμε τη συνεργασία μας με το Κοινοβούλιο για να αποφύγουμε την κατάσταση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και η συνεργασία αυτή δεν ε, χρησιμοποιήθηκε από την Κομισιόν. Σκοπεύετε να το κάνετε αυτό στο μέλλον. Επίσης για την αναθεώρηση της οδηγίας κοστιμάτων υπήρχε μια συζήτηση συγχωνεύσεων, επανεξετάσεων, αναθεωρήσεων. Δεν ξέρω αν οι οδηγίες αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τις αναθεωρούμε συνέχεια. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν έχουν εφαρμοστεί από κάποια κράτη-μέλη. Και τέλος, ε, ένα πιο προσωπικό σχόλιο. Την περασμένη φορά που ήσασταν εδώ και συζητήσαμε, σας ε, ρώτησα για το κυνήγι συγκεκριμένων πουλιών στη Μάλτα και τον περίοδο κυνηγιού την Ανησιάτικη Γιατί τοποθετήθηκε στην, στον κόκκινο κατάλογο από ένα εθνικό οργανισμό. Η Μάλτα έχει εξαιρέσεις βάσει της νομοθεσίας για την κυνηγετική περίοδο, αλλά εφόσον λαμβάνεται υπόψη το καθεστώς προστασίας των ειδών των συγκεκριμένων. Η Μάλκα λοιπόν παραβιάζει συγκεκριμένες αποφάσεις δικαστηρίου επ' αυτού, αλλά και την οδηγία του 2009 για την ποικιλότητα των τιμών και τις προσπάθειες ε, προστασίας των ειδών. Τι έχετε να πείτε για την κατάσταση αυτή και θα την αναφέρετε στην ανάληψη των δράσεών σας. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τζούντι Γκέρλιν, Ευχαριστώ και ευχαριστώ, Επίτροπε. Ευχαριστώ για την πληρέστατη παρουσίασή σας. Θα αναφερθώ στην ποικιλία της ατμόσφαιρας, όχι μόνο για το ενίσχυ e που τρέχει, αλλά με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το EIR, το οποίο αναφέρεται και το πώς αυτό θα λειτουργήσει. Γιατί μιλούμε για, το, για την ομοθεσία πλαίσιο, αλλά στην ουσία το σημαντικό είναι πώς θα εφαρμόζεται αυτή και θα επιβάλλεται. Έχουμε κυρώσει που εκκρεμούν κατά 16 κρατών μελών. Έχουμε καταδικαστικέ σε βάση του δικαστηρίου κατά ενό. Έχουμε ανάληψη δράση ε, κατά συγκεκριμένων κρατών, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία. Δεν είναι μικρά, μικρές χώρες αυτές. Έχουμε σοβαρά παραπτώματα. Και αναρωτιόμαι πώς αυτό θα λειτουργήσει στο πλαίσιο EIR. Γιατί θα έχουμε και μια έκθεση προόδου, αλλά το EIR θα εξετάσει πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε την επιβολή κυρώσεων και το να εξασφαλίσουμε ότι αυτές θα λειτουργούν και θα είναι απορρεπτικές. Γιατί εδώ μπροστά μας έχουμε την κατάσταση ότι οι κυρώσεις και οι παραβιάσεις αυτές είναι σχεδόν καθημερινές. Είναι μια καθημερινή πραγματικότητα και παρόλα αυτά δεν γίνεται καμία συζήτηση αποτροπή ή πρόληψης. Πώς λοιπόν θεωρείτε ότι θα λειτουργήσει το EIR ή στο πλαίσιο αυτό. Αναφερθήκατε στο φυσικό κεφάλαιο που είναι ένας ωραίος όρος. Είναι μια ωραία φράση. Εγώ στον Ηνωμένο Βασίλειο ε, ηγούμε μιας προσπάθειας ε, προτασίας των πουλιών, των τεινών. Ε, και ο κάθε οργανισμός που ασχολείται με την προστασία αυτή διαλέγει ένα συγκεκριμένο είδος. Εγώ επέλεξα, ο δικός μου οργανισμός επέλεξε ένα είδος που είναι παρόν σε 11 διαφορετικές χώρες επειδή μετακινείται και εκεί συζητήσαμε για τα οικοσυστήματα και, και κάποιες σοβαρότατες περιπτώσεις ε, κινδύνου που απειλείς για το είδος αυτό τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη δυστυχώ. και ε, καλό είναι όλο αυτό το ενδιαφέρον λοιπόν που εκφράζεται, αλλά πότε θα δούμε αποτελέσματα από αυτές τις προσπάθειες προστασίας. Ευχαριστώ κύριε Γερμπράντη για την άλλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς Επίτροπε που είστε εδώ και πάλι με μια ιδιαίτερα εμπιστευτομένη παρουσίαση. Τρεις ερωτήσεις να σας θέσω. Η πρώτη αφορά την εφορία εν γέννη. Όταν οριστικοποιήσαμε τους ε, στόχους της ε, του ΟΗΕ, αρχίσαμε να εξετάζουμε την επόμενη φάση. Εμείς, οικουμενικά παγκοσμίω, ε, είδαμε ότι η εξάλληψη της φτώχειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ακολουθήσουμε μία αηφόρο προσέγγιση. Γι' αυτό είχαμε και τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης. Πέρυσι στο Παρίσι αποφασίσαμε και συμφωνήσαμε ε, για συγκεκριμένου στόχου σε ό,τι αφορά την ε, οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι μόνο με τη βιώσιμη ανάπτυξη θα έχουμε την ανάπτυξη που θέλουμε και την οικονομική μεγέθυνση. Όμως, αν δει κανεί ε, τις ευρωπαϊκέ πολιτικές, όπω είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ή το Ταμείο του Γιούνκερ, το μόνο που λείπει είναι τα κριτήρια ε, βιωσιμότητας. Είχαμε στο παρελθόν ε, τέτοια κριτήρια που συνδέονταν με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αλλά πάνε πια αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την βιοπικιλότητα. Ε, παρουσιάσατε πέρσι την ενδιάμεση αναθεώρησή σας και τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά, ότι πρέπει δηλαδή επιγόντως να αναλάβουμε δράση ε, για να αλλάξουν τα πράγματα μέχρι το 2020. Αλλά από τότε δεν υπήρξε καμία συνέχεια. Απόλυτη σιωπή. Τι θα γίνει λοιπόν στου επιμέρου τομεί πολιτική, αλληλεία, θαλάσσια πολιτική κ.ο.κ. για να επιτύχουμε του στόχου μα. Και επίση για την βιοποικιλότητα. Ε, στο δάσο Βία βολέζα, το μόνο πρωτόγωνο δάσο που παραμένει στην Ευρώπη. Ε, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Γιατί η πολωνική κυβέρνηση ε, έχει στόχο να αρχίσει την υλοτόμηση σε αυτή την ε, πολύ σημαντική περιοχή. Και τέλο για την κυκλική οικονομία, Πρόεδρε. Παλαιότερα ήταν ζήτημα υψηλή προτεραιότητας σε πολιτικό επίπεδο μέχρι πέρσι, μετά την απόσυρση του παλαιότερου ε, πακέτου της δεσμημέτρων. Όμως τελικά βλέπουμε ότι ε, φεύγει το ενδιαφέρον και για τον οικολογικό σχεδιασμό υπήρχαν ε, υποσχέσεις και δεσμεύσεις, αλλά μόνο καθυστερήσεις βλέπουμε. Επομένω, παρακαλώ να διασφαλίσετε ότι θα παραμείνει ζήτημα υψή τη ε, προτεραιότητα η κυκλική οικονομία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Κονέτσινα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο τέλος ε, των σχολείων σας μας είπατε και πάλι ότι θέλετε να επικεντρωθείτε στην εφαρμογή των οδηγιών που έχουν ήδη υιοθετηθεί. Όμως, δύο χρόνια μετά την ακρόασή σα δεν βλέπω να έχει υπάρξει πρόοδος ε, στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Συνεχώς ε, θεσπίζεται και καινούργια νομοθεσία, κανονισμοί, οδηγίες, ενώ ξέρουμε ότι και η κείμενη νομοθεσία δεν εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη ε, πλήρως. Κάποιε φορές υπάρχουν και αντικειμενικοί λόγοι, άλλε φορές και για πολιτικούς λόγους. Κανείς δεν ακούει και δεν κάνουμε τίποτα. Εγώ θα προτιμούσα ε, να ξεκινήσουμε μια τάμπουλα ράσα, χωρίς, ε, αντί να ξεκινάμε με θέσπιση νέας νομοθεσίας που ξέρουμε ότι δεν θα εφαρμοστεί. Ιδίως σε ό,τι αφορά την ε, ποιότητα της ατμόσφαιρας, και πέραν της Τσεχίας βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες ε, που ρηπαίνουν, δεν ε, συμμορφούνται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αυτοί που πλήττονται τελικά είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ε, πολύ συχνά και σε γειτονικέ ε, χώρες, χωρίς να είμαστε σε θέση να κάνουμε κάτι και η Κομισιόν δεν αναλαμβάνει πραγματική δράση για να ε, αντιμετωπίσει το ζήτημα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, κάτι το οποίο δεν έχει αναφερθεί, αλλά είμαι βέβαιη ότι το παρακολουθείτε. οι εκπομπές που προκύπτουν από ε, τις ε, καλλιέργειες φινικελαίου βλέπουμε ότι έχουν προκύψει ακόμα και από χώρε όπως ε, η Γερμανία. Αλλά να μην επικεντρωθούμε μόνο σε εμά και στην Ευρώπη, αλλά και να δούμε τι θα κάνουμε για αυτά τα φαινόμενα. Γιατί βρισκόμαστε στο χείρο της καταστροφής και δεν υπάρχει η αντίστοιχη ανταπόκριση. θα περιορίσετε την χρήση φινικελαίου ιδίως από ε, καλλιέργειες που έχουν καεί. Θα υπάρξει νομοθεσία για την αποτροπή αυτού του φαινομένου. Και κατά δεύτερο λόγο, πώς ε, θα προσεγγίσετε τα βιοκαύσιμα, γιατί τα περισσότερα φινικέλαια αυτός, αυτή, αυτός είναι ο προορισμός τους, τα βιοκαύσιμα και είναι μια τεράστια αποτυχία, πρέπει να το περιορίσουμε. Ο Πρασίνος ο κύριος Όσλιν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία οικολογικής μεταστροφής της οικονομίας, αλλά όσον αφορά την βιοπικιλότητα, φαίνεται ότι, θα απο... ότι δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας για το 2020. Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση εξέδωσε πρόσφατα έκθεση. Από ό,τι φαίνεται δεν σημειώνουμε καθόλου πρόοδο. Και δεν βλέπω αντίδραση από πλευρά της Κομισιόν. Εάν αποτύχουμε και το 2020, τελικά καταλήγουμε να γίνουμε αναξιόπιστοι. Και αυτό συνδέεται και με την πολιτική γεωργίας μας. Έχουμε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Κάποιοι θέλουν ε, οικολογικό προσανατολισμό, αλλά άλλοι θέλουν ε, και πιο ε, ε, περισσότερη γεωργική εκμετάλλευση. Μήπως λοιπόν το greening, ο οικολογικός προσανατολισμός ε, τελικά αποδειχτεί σαπουνόφουσκα. Νομίζω ότι εάν δεν αλλάξουμε την γεωργική μας πολιτική θα αποτύχουμε. Και μία παρατήρηση ακόμα όσον αφορά τη γλυφοσάτη. Στην Γερμανία η αρμόδια αρχή λέει ότι η ουσία αυτή επηρεάζει αρνητικά την ε, βιοπικιλότητα, διότι σκοτώνει όλα τα φυτά. Γιατί δεν έχουμε ακούσει τίποτα από τη δική σας πλευρά για το θέμα αυτό. Και πού θέλετε να καταλήξετε όσον αφορά το Refit και το Natura 2000. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα του ελέγχου καταλληλότητας. Ποιος όμως ακριβώς είναι ο στόχος. Θα πείτε τελικά στι περιβαλλοντικέ οργανώσει ότι δεν έχει κανένα νόημα να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας. Μία προτελευταία ερώτηση. Όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού για τα λοιπάσματα. Εδώ και χρόνια στη Γερμανία δεν έχει γίνει σχετική αναθεώρηση. Ενώ η Κομισιόν ζητάει εδώ και χρόνια να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τι γίνεται λοιπόν στο θέμα αυτό και μία τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι θέλετε να βοηθήσετε όσον αφορά την ερμηνεία Πιστεύετε ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ε, θα πρέπει να έχουν ε, πρόσβαση ε, σε δικαστικές διαδικασίες, αλλά γιατί δεν δίνονται σχετικές εξηγήσεις στην ίδια την οδηγία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, Επίτροπε. Θα επικεντρωθώ στα δάση. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να περιορίσει την παράνομη κοπή των δέντρων η Κομισιόν και τα έσοδα από την παρανομικοποίηση αυτή και το εμπόριο και τη μεταποίηση. Θα πρέπει να έχουμε μια έλεγχο επίσης λέμε της προέλευσης του ξύλου. Ωστόσο στην Ευρώπη κυκλοφορούν σημαντικές ποσότητες ε, εισαγόμενου ξύλου υπόπτου προελεύσεως όπως λένε και οργανώσεις όπως η Greenpeace. Επίσης σχετικά με την ε, ανάχρηση της ε, αγροτικής γης ε, έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα σε σχέση με τα δάση. Δηλαδή δεν κόβουμε μόνο για το ξύλο αλλά κόβουμε για να έχουμε και παρθένο έδαφος για να το πούμε έτσι προς καλλιέργεια. Και εκεί καλλιεργούμε σόγια, φινικέλαιο, δέρματα, κρέας, την δηλαδή οι σόγια πάνε στη Γαλλία και στη Γερμανία, το δέρμα στην Ιταλία. Θέλω να πω όλε οι χώρε ε, καλύπτουν τα τρία τέταρτα των εισαγωγών αυτών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε παράνομα προϊόντα του δάσου ε, για ένα τζίρο άνω των 6 δι ετό. Είναι σαφέ ότι αν η Κομισιόν θα ήθελε να σταματήσει την αοψήλωση των δασών, θα, ήθελε και, θα έπρεπε και να περιορίσει αυτή την, ε, το εμπόριο αυτών των παράνομων ιδιών. Η παράνομη οψήλωση των δασών σύμφωνα με πρόσφατε μελέτε, ε, προκαλεί από μόνη της το 1 πέμπτο των συνολικών εκπομπών ε, ε, αερίων του θερμοκηπίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο μόνο ενόχο, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα από του πιο σημαντικού χρήστε παγκοσμίω. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να εφαρμόσουμε του ε, κανόνε πέραν του να κάνουμε ε, ελέγχου και στο πλαίσιο τη Συμφωνία των Παρισίων. Πώ εσεί θα αποτρέψετε λοιπόν παράνομα προϊόντα που προέρχονται από εδάφη που έχουν αψηλωθεί δάση. Σα ευχαριστώ. Προτού δώσω το λόγο στον Επίτροπο για απαντήσει. Έχουμε ακόμα 12 ομιλητές αργότερα και θα ζητήσω για το λόγο αυτόν από τον Επίτροπο να προσπαθήσει να κάνει μια προσπάθεια τουλάχιστον να περιορίσει λίγο τις απαντήσεις του. Σας ευχαριστώ Τζοβάνι. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Καρλ Χάιτς ε, Φλόρενς ε, για την στήριξη που δείχνει όπως πάντα. Ρώτησε λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό ο Καρλ για την πολιτική διαχείριση εμπορημάτων. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και επ' αυτού να αποδώσουν καλύτερα. Καταρχά η ιδέα του στόχου τη θέσπιση στόχων δεν είναι μόνο προ την κατεύθυνση των κυρώσεων αλλά και προ την κατεύθυνση τη καλύτερη παρακολούθηση και επιτήρηση των κρατών μελών προκειμένου εκείνα να βελτιώσουν την επίδοσή του, γιατί είναι τα κράτη-μέλη στο τέλο που θα επωφελούνται περιβαλλοντικά και οικονομικά από την ε, καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων και μετατροπή τους σε πόρο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πρώτα απ' όλα, όπου θα εντομίζουμε κενά από μια πρώιμη ήδη φάση για να μπορούμε να αναλαμβάνουμε δράση ήδη πολύ νωρί. Επίσης προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη μέσω τεχνικών συμβουλών, επιβελτίστων πρακτικών επί περιοχών ή στις οποίες θα έπρεπε να επενδύσουν περισσότερο. Πέρα από τις τεχνικές αυτές συμβουλές, διαθέτουμε και χρηματοδοτική στήριξη, κυρίως μέσω του ορίζοντα 2020, η IB, διαθετικά ταμεία κτλ. Μόνο επί της διαχείρισης απορριμμάτων θα διατίθενται περί τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο, μόνο για αυτά τα έργα από τώρα και μέχρι το 2020. Βεβαίως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε τι πλαίσιο θα χρησιμοποιούνται οι πόροι αυτοί. Όταν μιλούμε για διαχείριση απορριμμάτων δεν θέλουμε στην κάτω κλίμακα της ιεραρχίας της διαδικασίας αυτής θέλουμε να επενδύσουμε στην επανάχρηση των γεών και θέλουμε να κινηθούμε και στην καύση, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που θα συζητηθεί περίπτωση προς περίπτωση. Έχετε δίκιο ότι για τα κράτη-μέλη δεν έχουν καν ξεκινήσει. Είναι αλήθεια. Και αυτό είναι αλήθεια, αν θέλετε, σε όλο το φάσμα της δραστηριότητα. Έχουμε 28 κράτη-μέλη που παρόλο έχουμε την ίδια νομοθεσία, τους ίδιους στόχους, τα 28 αυτά κράτη κινούνται σε 28 διαφορετικές ταχύτητες. Μερικές φορές χρειάζεται μαστίγιο και μερικές φορές χρειάζεται καρότο. Και έπρεπε και να προωθούμε και να υποστηρίζουμε. Να ενισχύουμε και να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη. Μιλήσατε για τα χωροκατακτητικά είδη. Αυτό που κάναμε όπως γνωρίζετε είναι ότι καταρτήσαμε τον κατάλογο των ειδών αυτών για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν τρία είδη παρεμβάσεων. Πρόληψη, έγκαιρη, έγκαιρος εντοπισμός και AIS. Ο κατάλογος δηλαδή. Ο οποίος έλαβε πολύ θετική άποψη από την ε, Επιτροπή το Δεκέμβριο πέρυσι αλλά δεν ενεκρίθη διότι έφερε αντίρρηση το Κοινοβούλιο ότι η Κομισιόν είχε υπέρβαση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της. Ιδιαίτερα για συγκεκριμένα είδη του καταλόγου όπως το ρακούν, αλλά και η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει την πρώτη επικαιροποίηση του καταλόγου αυτού. Και αυτό που θέλω κυρίως να πω είναι ότι αυτός ο κατάλογος είναι καρπός επιστημονικής μελέτης και προσέγγισης, συνάδει και συμμορφούνται προς τον κανονισμό και θα επικαιροποιούμε τον κατάλογο αυτό όπως απαιτεί και η AIS για το ανεξιάτικο κυνήγι στη Μάλτα. Και εγώ ανησυχώ. Και θα σας πω ότι εγώ ζήτησα από τις υπηρεσίες μας να αναλάβουν δρέση σε αυτό. Οι αρχές της Μάλτας έχουν ήδη κληθεί να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Τους εδόθησαν 10 μέρες. Όπως λοιπόν αναλάβαμε δράση και σε προηγούμενες περιπτώσεις στη Μάλτα για το κυνήγι συγκεκριμένων πουλιών, θα το ξανακάνω. Και θα το ξανακάνουμε. Πρέπει να δούμε κατά πόσον η εξαίρεση που χρησιμοποιεί η Μάλτα ευθυγραμμίζεται προς την οδηγία ή όχι. Οι εξαιρέσεις. Για το fitness check. Και για να απαντήσω και στην Τζούλια που αναφέρθηκε στο fitness check και στη βιοπικιλότητα. Να πω πρώτα απ' όλα ότι για το check η Κομισιόν προχωρεί. Δεν μείναμε μόνο στην υλοποίηση την αρχική, ε, ερευνούμε ακόμα αποκλήσεις και παραβιάσεις και μπορώ να μιλήσω όχι για συμπεράσματα αλλά για πρώτες ενδείξεις που έχουν απτυχθεί από συμβούλους εξωτερικούς, όχι της, εσωτερικά της Κομισιόν. Οι ενδείξεις λοιπόν που έχουμε είναι ότι πρέπει να χρεια... ότι χρειαζόμαστε παραλαμβάνω μιλούμε για ενδείξεις αλλά φαίνεται ότι δεν χρειάζεται να ανοίξουμε συζήτηση για άλλο fitness check ότι χρειαζόμαστε υλοποίηση και εφαρμογή ωστόσο εγώ έχω τις ανησυχίες μου διότι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν θέλουν να ενισχύσουν το πλαίσιο βιοπικιλότητα θα είναι οι πρώτοι που θα επικρίνουν ότι δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας το έτος 2020. Δηλαδή και να ανοίξουμε το πακέτο και να μην το ανοίξουμε όπως και να γίνει θα χρειαστεί να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιτύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει για το 2020. Εγώ παραπέμπω στην έκθεση της, του, της κατάστασης ε, στη φύση, στη βιοποικιλότητα και στο περιβάλλον, αυτές οι εκθέσεις τι λένε. Λένε ότι έχει επιτευχθεί κάποια, κάποια πρόοδος. Ωστόσο έχουμε σαφέστατες και ξεκάθαρες ενδείξεις ότι δεν θα επιτύχουμε, δεν θα καλύψουμε τους στόχους μας μέχρι το 2020. Και δεν θα έχουμε Ενδιάμεσε εκθέσεις του 2020, θα είναι τελικές εκθέσεις. Επιτύχαμε ή όχι. Ή τσεκ ή χ θα έχει η έκθεση. Ή πράσινο ή κόκκινο. Κάποιος από εσάς αναφέρθηκε στην ε, Γεωργία. Έξω έχω παράδειγμα. Όλες οι εκθέσεις αναφέρουν τη γεωργία ως μία από τις βασικότερες αιτίες της έλλειψης της απώλειας βιοποικιλότητας. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να ενισχύσουμε το πλαίσιο της νομοθεσίας της οδηγίας μας. Θα αναφερθώ στη Γεωργία αργότερα, όχι στο σύνολο της. Εγώ μπορώ να ασκήσω κριτική για πρακτικές που δεν είναι καλές, που συμβαίνουν στο, στο πεδίο της γεωργίας, αλλά υπάρχουν και καλές πρακτικές. Για το πλαίσιο. Ξέρετε ότι αυτό ήταν ένα εγχείρημα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την συλλογή δεδομένων, την υποβολή εκθέσεων. Είχαμε ακόμα και κάποιες ε, διαβρυντικέ ε, αποστολέ σε ορισμένα κρατημέλη και ουσιαστικά ο σκοπό μα είναι μια αξιολόγηση σε πέντε κατηγορίε. Θέλαμε να δούμε την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνοχή, ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία και συνάφεια αυτών των οδηγιών. Όπως γνωρίζετε όλοι, είχαμε πάνω από μισό εκατομμύριο απαντήσεις, 550.000 απαντήσεις, πολύ περισσότερες ε, από ό,τι στο TTIP. Και τα ευρήματα συζητήθηκαν πέρσι τον Νοέμβριο στις Βρυξέλλες. Το σχέδιο έκθεσης το λάβαμε τον Φεβρουάριο του 2016 και στις αρχές του Ιουνίου θα έχουμε την παρουσίαση των ε, αποτελεσμάτων. Και τότε βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει συνέχεια στο φετινό εγχείρημα. Η Τζούλη επίσης μίλησε ε, για ορισμένα είδη πουλιών στο Ερμηνο Βασίλειο. Το έχουμε συζητήσει και Ε, Ναι, ανησυχώ. Όντω, οι κυνηγοί σκοτώνουν πουλιά, συμβαίνουν όλα αυτά. Όμω, έχουμε και γεωργικέ πρακτικέ, ε, λοιπάσματα, ζανιοκτόνα, κλιματική αλλαγή. Και όλα αυτά σκοτώνουν επίση ε, τα πουλιά. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε για αυτή τη συζήτηση. Πρέπει όλα αυτά να τα εξετάζουμε παράλληλα. Και σίγουρα θα έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε, γιατί τελικά κύριος ε, στόχος μας είναι ένας, να σώσουμε τα πουλιά και τη βιοποικιλότητά μας. Ο κύριος Γερμπράντη μίλησε για την βιωσιμότητα και συμφωνώ απολύτως. Αν δείτε και το έργο μας, ε, τη ρητορική μας για τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, όλα αυτά συνδέονται με τη βιωσιμότητα, την αηφορία, και μιλήσατε και για την οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα και εγώ προωθώ την προτεραιότητα για την ε, διακυβέρνηση των ωκεανών και ούτω καθεξής, γιατί κάτι που δεν κατάλαβα όταν μιλήσαμε για την κλιματική αλλαγή και την ε, οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, δεν εξετάσαμε σχεδόν καθόλου το ζήτημα των ωκεανών. Μόνο σε μία εκδήλωση στο περιθώριο της COP21 ε, εξετάσαμε το ζήτημα των ωκεανών. Ενώ γνωρίζουμε ότι έχουν τεράστια συμβολή σε ό,τι αφορά ε, το διεξίδιο του άνθρακα οι ωκεανοί στο πλανήτη μας. Για την βιοπικιλότητα, όντως, και πάλι θέλουμε κάτι περισσότερο από την ενδιάμεση αναθεώρηση. Χρειαζόμαστε ενέργειες που ακολουθούν την ενδιάμεση αναθεώρηση για να δούμε πόσο επιτυχάνονται οι στόχοι 2020. Προφανώς υπάρχουν ε, διάφορες ε, πολιτικές ε, προσεγγίσεις. Έχουμε το fitness check, συζητήσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, εφαρμογή των στόχων, ε, των αναπτυξιακών στόχων της χειρετηρίδας και μάλιστα των βιώσιμων στόχων αυτών. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει, τους έχουμε προσυπογράψει, όμως το πιο σημαντικό είναι να τους εφαρμόσουμε κιόλα. Σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία, είμαστε 100% βέβαιοι ότι η κυκλική οικονομία παραμένει ε, ανάμεσα στις πρώτες ε, προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό ισχύει. Είναι ε, μία δέσμευση του Σώματος των Επιτρόπων. Και ο Γίγκη Κατάινεν πριν από μερικές ημέρες την ίδια διαβεβαίωση σας έδωσε. Για αυτό το δάσος στην Πολωνία που αναφέρατε, όντως και εμάς μας προβληματίζει αυτό το ζήτημα. Και μας προβληματίζει όχι μόνο το ότι πρόκειται για έναν μοναδικό ε, χώρο που προστατεύεται από το Natura, αλλά και από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Και θέλουμε να αποφύγουμε ε, βλάβες που δεν μπορούν να θυρωθούν στο μέλλον εάν ε, εφαρμοστούν όντως αυτές οι αποφάσεις ε, υλοτόμησης σε αυτό το δάσος. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο και ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στο δάσος θα συνάδει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Για να ξέρετε, έχουμε ήδη ξεκινήσει έναν ευρωπαϊκό πιλότο, ε, ένα πιλωτικό πρόγραμμα τώρα τον Απρίλιο και Κατόπιν διαβούλευση με τι πολωνικέ αρχέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει ποια θα είναι η επόμενη ενεργειά τη. Ο κύριος Γκεμπράντη επίσης ε, μίλησε για τον οικολογικό σχεδιασμό και προετοιμάζεται ε, το νέο πρόγραμμα οικολογικού σχεδιασμού και αυτό εντάσσεται, όπω ξέρετε, στο πρόγραμμα εργασιών μα. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των οδηγιών και το EIR. Πρόκειται για ένα πολύ καλό εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει να συνδράμουμε τα κρατημέλη και από πού προκύπτει αυτή η πρόταση, από το ότι έχουμε τέτοιες ε, ειδικέ αναχώρα εκθέσεις σε πολλούς διαφορετικούς τομείς πολιτικής. Γιατί να μην κάνουμε το ίδιο και για το περιβάλλον. Ούτως ώστε κάθε κράτος μέλος να έχει και μια αναθεώρηση των επιδόσεών του. Σκοπός είναι λοιπόν να συζητήσουμε από κοινού με τα κρατημέλη ποια είναι τα προβλήματα, η ε, στενοπή και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τυχόν προβλήματα. Βεβαίως και θα ενημερώνουμε και το Κοινοβούλιο και ε, θέλουμε να κάνουμε ανατατά χρονικά διαστήματα να υποβάλουμε εκθέσεις. Για το φινικέλαιο. Γνωρίζω ότι οι περισσότεροι ευρωβουλευτέ θεωρούν ότι το φινικέλιο θα πρέπει να απαγορευτεί εξαιτία τη αποψήλωση ε, των δασών που θεωρείται ότι προκαλεί. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει διακρίσει μεταξύ των φυτικών ελαίων. Γνωρίζουμε ότι το φινικέλαιο είναι σημαντική πηγή εισοδήματο και απασχόληση στι περισσότερε χώρε παραγωγού. Όμω έχουμε ε, και είναι σημαντική ανησυχία ότι μπορεί να ενδεχομένω να ζημιώνει και ε, να βλάπτει οικοσυστήματα και ζωικά είδη. Γι' αυτό θέλουμε από κοινού ε, με τις χώρες παραγωγούς να εξετάσουμε πώς μπορούμε να ε, περιορίσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο και να ενθαρρύνουμε ή ακόμα και να στηρίξουμε οικονομικά άλλες μεθόδους και πιο βιώσιμη παραγωγή. Έχουμε εξετάσει βεβαίω και το θέμα τη αποψήλωση. Η Κομισιόν συνεχώ ε, εξετάζει πώ μπορούμε να εντείνουμε τη δράση μα ε, κατά τη αποψήλωση και υποβάθμιση των δασών. Για την ε, βιοπικιλότητα, νομίζω ήδη το θίξαμε νομίζω, η γεωργική πολιτική, ναι, είναι κάτι που με προβληματίζει ιδιαίτερος και εδώ χρειάζομαι και τη δική σας στήριξη. Ιδίω με ό,τι αφορά και την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Ε, δεν ξέρω, ίσω και στη δεύτερη παρέμβασή μου θα μπορούσα να απαντήσω άλλα τέτοια ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να σκεφτούμε τώρα ότι έχουμε 12 ομιλητές και θα πρέπει να απαντήσει και ο Επίτροπος και μας ε, Μένουν 15 λεπτά. Θα πρέπει λοιπόν να στήσω από του ομιλητέ να είναι πάρα πολύ σύντομοι. Δίνω το λόγο πρώτα στον Ιβο Μπέλετ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα περιοριστώ σε μία ερώτηση. Επίτροπε, εδώ μπροστά σα βρίσκομαι. Μία ερώτηση. Αναφερθήκατε στην ποιότητα του αέρα. Και η ερώτησή μου είναι όσον αφορά τα μικροσωματίδια και ιδιαίτερα όσον αφορά τη θέρμανση των κατοικιών. Οι υπολογισμοί από γνωστά Ινστιτούτα δείχνουν ότι το 15 έως 21% των μικροσωματιδίων προέρχονται από την θέρμανση κατοικιών που γίνεται κυρίως με ξύλα και άνθρακα. Έχουμε υιοθετήσει κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού για την θέρμανση, αλλά τα κριτήρια αυτά θα τεθούν σε ισχύ από το 2022. Στο μεταξύ, αρκετά κράτη-μέλη έχουν ήδη εφαρμόσει πιο αυστηρούς κανόνες, έχουν ξεκινήσει εκστρατείες ε, και έχουν δώσει οικονομικά κίνητρα στον κόσμο να αλλάξει ε, τον τρόπο θέρμανσης ε, της κατοικίας του. Δεν θεωρείτε λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο να προωθήσουμε πιο γρήγορα την χρήση πιο καθαρών θερμαστρών να δώσουμε κίνητρα δηλαδή για την αντικατάσταση των ε, των συστημάτων θέρμανσης κατοικιών που γίνεται με τόσο μη αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Ποναφέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά σας, καθώς και για την συνεργασία που είχαμε ε, όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για τα απόβλητα και θα ήθελα να συζητήσω το θέμα αυτό μαζί σας τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπατε, υπέβαλε πρόταση για την αναθεώρηση της νομοθεσίας του κανονισμού για τα λοιπάσματα και έχουμε επίσης το θέμα του οικολογικού σχεδιασμού. Η πρόταση λοιπόν για τον ε, κανονισμό λοιπασμάτων αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για την κυκλική οικονομία, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ε, βιολογικά απόβλητα για να ε, προωθήσουμε την οικονομία μας. Ωστόσο, πιστεύω ότι δεν καλύπτεται επαρκώς η σχέση ανάμεσα στα βιοδιασπόμενα πλαστικά και την δυνατότητα χρήσης τους ως λιπάσματα. Ξέρω ότι αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και μάλιστα έχει προταθεί από μια σειρά κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε το θέμα αυτό, ωστόσο αποφάσισε να μην το συμπεριλάβει στην συγκεκριμένη πρόταση, αλλά σε πρόταση για τα πλαστικά το 2017. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς έχουν τα πράγματα και ποια είναι η στρατηγική για τα πλαστικά θα έχουμε τη δυνατότητα να αρχίσουμε να ε, ασχολούμαστε με άλλες προτάσεις. Ξέρω ότι είναι ε, πολύπλοκο το θέμα, διότι μόνο το 20% των πλαστικών ανακυκλώνεται αυτή τη στιγμή. Τι θα μπορέσουμε να κάνουμε για να πετύχουμε τους στόχους ανακύκλωσης που προβλέπονται στο νέο πακέτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζουίτεμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ. Έχω ε, μία ερώτηση όσον αφορά τον έλεγχο καταλληλότητας για την οδηγία για τα πτηνά. Είπατε ότι έγινε πολύ καλή διαβούλευση, πάνω από 500 ε, απαντήσεις ελήφθησαν. Γνωρίζετε όμως ότι πολλές από τις απαντήσεις αυτές ε, εστάλησαν σε έντυπο στο διαδίκτυο και ότι κάποια ομάδα ενδιαφερομένων ε, ξεκίνησε μεγάλη εκστρατεία ώστε ο κόσμος να συμπληρώσει τα έντυπα αυτά και να σας τα στείλει. Θεωρείτε λοιπόν ότι με την αποστολή αυτών των εντύπων μπορεί να στρεβλωθεί η εικόνα και αυτό έχει ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των συστάσεων, διότι ελπίζω ότι στο πλαίσιο των συστάσεων θα υπάρχει χώρος για καινοτόμες και πραγματικές λύσεις και για νέες γνώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίζεκε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για την εκτενή εισαγωγή σας και για την συζήτηση. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με την σχέση περιβαλλοντικής πολιτικής και πολιτικής αλληλείας. Αναφέρομαι κυρίως ε, στην αλληλεία στη Βόρεια Θάλασσα. Ε, είχαμε ήδη αναφερθεί στο θέμα αυτό. Το 2015 και έχουν δοθεί 13 άδειες ε, στην ε, Γερμανία και στην Ολλανδία περισσότερες ε, για πιλωτικό πρόγραμμα και μέχρι το καλοκαίρι του 2015 θα έπρεπε να έχουμε την έκθεση αξιολόγησης, αλλά πλησιάζει το καλοκαίρι του 2016 και δεν έχουμε σχετική έκθεση Πάντως ε, σε ειδικό περιοδικό των κάτω χωρών ε, φαίνεται ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα αυτή η ε, αλληλεία με ηλεκτρισμό και το θέμα είναι τι θα πρέπει να γίνει. Ε, θα ήθελα πολύ να γνωρίζω. Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σκοτοκρότε. ευχαριστώ. Μόλις συζητήσαμε τι δεν λειτουργεί πολύ καλά, τι δεν είναι ιδιαίτερα θετικό, αλλά συχνά όταν μιλάμε για την προστασία ειδών ε, βλέπουμε υπερβολική επιτυχία. Για παράδειγμα κάποιες χήνες ε, στην ε, κάτω Σαξονία. υπάρχουν μέτρα μέχρι 31 Τρίτου όσον αφορά το κυνήγι, αλλά με ε, την αλλαγή του κλίματος έχουν αλλάξει οι εποχές και έτσι τώρα πια έχουμε χιλιάδες ε, τέτοιες χήνες οι οποίες ε, βρίσκουν ζωοτροφή στα λιβάδια και ε, έτσι καταστρέφεται μεγάλο μέρος της φύσης από αυτήν την ασπρομαγουλόχυνα. Και θα πρέπει να βρούμε μία λύση με φυσικό τρόπο, για παράδειγμα την αφαίρεση των αυγών, ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε για τη δυνατότητα της σημερινής συζήτησης. Δύο ερωτήσεις έχω. Αναφερθήκατε ε, στον Ιδράργυρο και την ε, Σύμβαση Μιναμάτα. Είμαι η συγητής για την έκθεση αυτή και θα ήθελα να θέσω την ε, ερώτηση εάν τα σφραγίσματα στα δόντια θεωρείται ότι είναι ύποπτα όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία. Ξέρετε, τα παιδιά όταν τρώνε πολλό γλυκά παίρνουν σφραγίσματα. Και επίσης βλέπουμε μεγάλη απώλεια της βιοπικιλότητας. Και αυτό γίνεται κυρίως για να καλλιεργηθούν ε, ζωοτροφές ε, για να διασφαλίσουμε δηλαδή την παραγωγή κρέατος ε, που έχει όμως πολλές αρνητικές συνέπειες σε πολλούς άλλους τομείς. Βλέπουμε μόνο καλλιέργειες και Σύντομα, πρόσφατα συγγνώμη, η κινέζικη κυβέρνηση ανακοίνωσε πολύ φιλόδοξο στόχο να μειώσει την κατανάλωση κρέατος στην Κίνα κατά 30% μέσα στα επόμενα 15 χρόνια για να αντιμετωπιστεί η αλλαγή του κλίματος. Η ερώτησή μου κύριε Βέλα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πότε θα προχωρήσει σε μείωση της παραγωγής του κρέατος ή είναι τελείως ταμπού το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mr. Σας ευχαριστώ κύριος Φρόντε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Να θυμίσω ότι για την εισαγωγή προϊόντων ξυλίας ε, παράνομης κοπής δεν έλαβα απάντηση. Θα ήθελα να λάβω μια απάντηση. Για τα στόκ ε, των ε, τα αλλιευτικά. Ε, είχαμε συναντηθεί στην Κατάνια επί του θέματος αυτού και ξαναείδαμε την κατάσταση είδαμε ότι είναι πολύ σοβαρός ο αντίκτυπος και ο κλιματικός και ο περιβαλλοντικός και ο της μολύνσεως και της ρήπανσης. Δεδομένων όλων αυτών, καθότι βρισκόμαστε σε μια ανισχυτική λοιπόν κατάσταση, όλοι περίμεναν μια απάντηση της Κομισιόν προκειμένου να καταλάβουν πώς τελικά θα παρεμβαίναμε στα αλληλευτικά αποθέματα ώστε να τα αποκαταστήσουμε το 90% των αποθεμάτων είναι υπεραλλιευμένα. Έχετε κάποιο input από πλευράς κομισιών για να καταλάβουμε τι θα κάνουμε σχετικά με αυτά τα οικοσυστήματα και αυτά τα αποθέματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μέλιορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω σε μια ερώτηση, κύριε Επίτροπε, και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με αυτό που ανέφερε ήδη ο κύριος Χόισλινγκ. Γεωργική πολιτική και βιοπικιλότητα. Εσείς είπατε πριν ότι το 80% των εκτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκτάσεις δασικές και γεωργικές. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα τι πρέπει να γίνει καλύτερα στην γεωργία ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας ε, περί βιοπικιλότητας για το 2020 για να μπορούμε να πλησιάσουμε τους στόχους μας ε, και όσον αφορά τον έλεγχο καταλληλότητας της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής βλέπουμε ότι το greening, ο οικολογικός προσανατολισμός υποτίθεται ότι θα ήταν το η λύση για όλα, αλλά δεν λειτουργεί πολύ καλά. Μήπως λοιπόν μπορούμε να πετύχουμε με κάποιο τρόπο περισσότερη πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Περίκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα... Εδώ κάθομαι. Θα ήθελα να ακουστεί και κάτι διαφορετικό για τον έλεγχο καταλληλότητα. Συμφωνώ με τον κύριο Χέτεμα, αλλά το έχω πει ξανά και ξανά ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα και σχόλια επιχειρήσεων που ε, δεν εισακούονται και θα σας δώσω και ορισμένα παραδείγματα. Έχουμε το διάφορα πάρκα Natura, τα οποία είναι πολύ σημαντικά Όμω έχουμε παράλληλα και συγκεκριμένου καλλιεργητέ που δεν μπορούν να κρατήσουν τις καλλιέργειέ τους γιατί δεν μπορούν να κόψουν καν τα δέντρα πάνω στι καλλιεργίες του. Μετά πώς μπορεί κάποιος ε, ε, να αποδείξει ότι υπάρχουν ε, ζημίες. Μετά στη δική μου περιοχή και στρέφουμε και στον κύριο Καρλ Άιντ Φλόρενς, ότι πλήττονται συγκεκριμένοι γεωργοί παρότι προσπαθούν ε, να διατηρήσουν το περιβάλλον εδώ και χρόνια. Πολλά παραδείγματα μπορώ να φέρω, αλλά ποια είναι η λύση. Υπεψηφίσαμε το ψήφισμα για τον ιό Ζήκα. Ναι, να καταπολεμήσουμε τον ιό, αλλά μαζί με την πρόληψη πρέπει να λειτουργήσουμε, κύριε Επιτροπέ. Τι γίνεται με τους αντίστοιχους ε, βιοτόπους ε, Natura. Κατά τη γνώμη δεν έχει υπάρξει κατάλληλη αντιμετώπιση, γιατί νομίζω ότι δεν λειτουργείται αμερόληπτα. Και τέλος, και οι γεωργοί είναι αυτοί που ε, προσπαθούν να προστατεύσουν στο περιβάλλον, αλλά εξαφανίζονται. Ο κύριος Θορίνιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για, τον, για την πληρέστατη και σαφέστατη παρουσίασή του. Ήσασταν πολύ σαφή σχετικά με τους στόχους που πρέπει να έχουμε στο θεματολόγιο. Όπως είπε και ο Επίτροπος, προκειμένου να εφαρμόσουμε, να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς και επιθυμούμε να έχουμε εφαρμογή και υλοποίηση, χρειαζόμαστε να πλησιάσουμε τους πολίτες και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα δέσμευσης, δεσμεύσεων και εμπιστοσύνης. Αναφερόμενος ε, λοιπόν στις ε, πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ασφαλείας η Κομισιόν υπέβαλε ένα ενδεικτικό πυρηνικό πρόγραμμα το οποίο είναι τελείως εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή μόνο για να είμαστε μέσα στους στόχους του 2020 θα πρέπει να καταργήσουμε, να κλείσουμε όλες σχεδόν τις πυρηνικές μας ε, εγκαταστάσεις. <coughs> Χρειαζόμαστε εκτεταμένους πόρους που δεν έχουμε διαθεσή μας. Η Ισπανία, για να φέρω ένα άλλο παράδειγμα, θα χρειαστεί να επενδύσει 15 δισεκατομμύρια σε πόρους προκειμένου να επικαιροποιήσει τις δικέ τη εγκαταστάσει. Υπάρχουν επίσης κρούσματα, ατυχήματα μικρής έκτασης αλλά και ε, ε, πιο σημαντικής έκτασης επιμολύνσεων, ποταμών κτλ. Εδώ λοιπόν, ακριβώς σε αυτό το σημείο έχουμε τον θεμελιώδη λίθο της ε, έδρασης της εμπιστοσύνης με τους που πρέπει να έχουμε να επιτύχουμε από τους πολίτες. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Επιτροπή, για τις απαντήσεις σας. Λοιπόν, ο κύριος Αφρόντε αναφέρθηκε στην ε, παράνομη ξυλία και τα αντίστοιχα προϊόντα έχουμε, το γνωρίζουμε το πρόβλημα και έχουμε προβλήματα και με συγκεκριμένε τρίτες χώρε αλλά και εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ήδη αναλάβει δράση για παραβιάσεις από πλευρά συγκεκριμένων κρατών μελών. Ο Ήβο μίλησε για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που το έχουμε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κορυφώνεται σε συγκεκριμενα κρατημέλη δεν θα έλεγα σε πολλά, αλλά δύο από αυτά τα κρατημέλη που εγώ επισκέφθηκα ανέλαβαν λεπτομερείς και, και εξαντλητικές συζητήσεις. Εστιαζόμαστε λοιπόν μαζί με τα κρατημέλη στα συγκεκριμένα αυτά προβλήματα και στον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για τα λοιπάσματα που αναφέρθηκε η Σιμώνα, η κυρία Μποναφέ. Η αναθεώρηση των οδηγιών και η συνεισφορά του στην κυκλική οικονομία είναι προφανής. Αλλά βιοποικιλότητα σημαίνει και καλύτερη χρήση και χρησιμοποίηση των πόρων. Κάτι τέτοιο θα βελτίωνε και την υγεία του υπεδάφους αλλά και η αντικατάσταση θα έπρεπε να γίνει των λοιπασμάτων που εις στο άζωτο. Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει εκτενώς σχετικά με τον κύκλο ζωής των προϊόντων αυτών, την ετικετοθεσία και χωρίς η μόρφωση προς τις προϋποθέσεις αυτές ε, δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν αυτά τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ ε, θα ξανααναφέρω το θέμα των ε, λιπασμάτων με μητρώδη. Τώρα για τα πλαστικά. Είχαμε στο σχέδιο δράσης ε, αναπτύξει μια στρατηγική για τα πλαστικά. Ήδη από το 2013 είχαμε ένα έγγραφο σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων πλαστικών και υπήρχε και ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Είχε λοιπόν τεθεί ένα πλαίσιο στρατηγικής με ευρία διαβούλευση και η πράσινη βίβλο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο περαιτέρω σχεδιασμό της στρατηγικής αυτής. Τώρα βέβαια κάποια σημεία του ψηφίσματος τα έχουμε ήδη ενσωματώσει και τα υλοποιούμε ήδη όπως την σταδιακή απόσυρση των χωματερών και την ανακύκλωση των πλαστικών. Για την ε, βιοχημική διαχείριση των πλαστικών λιπασμάτων έχει ζητήσει η Κομισιόν την άποψη ε, εξωτερικών συμβούλων Θα έχουμε τα αποτελέσματα των μελετών αυτών, ελπίζω, μετά το καλοκαίρι, σχετικά με τη βιοδιάσπαση, τη βιοδιασπασιμότητα μάλλον των υλικών αυτών, το οποίο αφορά και στη συζήτηση των θαλασσών και της ε, θαλάσσιας ρήπανσης. Ο κ. Γουιτέμα αναφέρθηκε στο Βίνες Τσέκ, αν θα πρέπει να δούμε ως αυτές τις 550.000 ε, απαντήσεις ως απαντήσεις χωριστές μεταξύ τους ή ως ένα ενιαίο επιχείρημα. Το γεγονός ότι έχουμε 550.000 απαντήσεις σημαίνει ότι είναι ανησυχίες που εκφράζουν 550.000. Και είχαμε βεβαίως κράτη-μέλη, μη όμικρον, ειχαμε είχαμε επιστολές υπουργών από διάφορα κράτη-μέλη, είχαμε γεωργούς, κυνηγού, δασονόμους. Όλα αυτά εξετάστηκαν από, την, ε, από τους συμβούλους και λύθησαν υπόψη. Ε, Γκίζεκε. αυτές οι συγκεκριμένες τεχνικές αλληλείας ε, που χρησιμοποιούνται στη Βόρεια Θάλασσα, που χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό ρεύμα. Πρόκειται για μια νέα τεχνολογία και σε πρώτη ανάγνωση περιορίζουν τα παραλίευματα γιατί είναι πιο στοχευμένες και μάλλον μολύνουν λιγότερο τον πυθμένα των θαλασσών. Όμως, ακόμα δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με αυτό δεν κατανοούμε απολύτως όλα τα συστατικά, της λεπτομέρειες του οικολογικού αντικτύπου της μεθόδου αυτής. Δηλαδή υπήρχε ένα επιχείρημα ότι όταν βυθίσουμε ηλεκτρικά φορτισμένα καλώδια μπορεί κάποιο είδος να μην παγιδευτεί αλλά να υποστεί ανεπανόρθωτη σωματική βλάβη. Εκεί χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερες επιστημονικές ενδείξεις. Υπάρχει, υπάρχουν κάποια σκάφη που έχουν ενταχθεί σε ένα πενταετές πρόγραμμα αλίας με ηλεκτρικό παλμό, εν πάση περιπτώσει, με ηλεκτρικό φορτίο, Προς το παρόν προσπαθούμε να συλλέξουμε τις ενδιάμεσες εκθέσεις για τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να έχουμε πληρέστερη εικόνα. Αλλά δεν βασιζόμαστε μόνο σε αυτήν. Είχαμε και πρόσφατες αποστολές συλλογής δεδομένων σε Ολλανδία και Γερμανία μεταξύ άλλων για να δούμε πώς επιθεωρούν, επιτηρούν, ελέγχουν την μέθοδο αυτή αλίευσης τα κράτη και έχουμε ζητήσει από τα κράτη αυτά να αναλάβουν συγκεκριμένα μέτρα, θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε και να επιτηρούμε. Όχι μόνο την ίδια τη διαδικασία, αλλά και την, τις εξελίξεις που θα έχουμε στις αλληλευτικές ζώνες και στο οικοσύστημα. Ο κύριος Γκρότε, ναι, υπάρχει ένα ζήτημα. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη έχουν το πρόβλημα αυτό με, με, με χήνες ε, σε κάποια κράτη-μέλη, με, με λύκους σε κάποιες άλλες ε, περιπτώσεις, ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη. Πρέπει κανείς να έχει μια ισορροπημένη και συνολική προσέγγιση. Κάποιες φορές νομίζω ότι παρασυρώμαστε ε, για να μην για να, προστα... για να υπερπροστατεύσουμε ένα είδος ή για να κάνουμε ακριβώς το αντίστροφο. Προσπαθούμε να βρούμε μια φυσική ισορροπία. Και παρότι λησμόνησα να αναφέρω την Natura 2000, αν, αν δούμε τις περιοχές Natura 2000 και τις εξετάσουμε, βλέπουμε πολύ μεγάλη πρόοδο. σε εκείνε τουλάχιστον περιοχέ που υφίστανται μια πλήρη και αποτελεσματική διαχείριση. Όχι τι άλλε. Επομένω δεν μα αρκεί να, κα... να ταυτοποιήσουμε τι περιοχές Natura 2000 αλλά και τη διαχείρισή του. Αναφερθεί και στον Ιδράργυρο. Ναι. Η επικύρωση τη σύμβαση Μιναμάτα θα είναι υποφελή για όλου υπό την περιβαλλοντική σκοπιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και 26 κράτη-μέλη υπέγραψαν μαζί με 100 άλλα κράτη τον Οκτώβριο του 2014 αλλά προκειμένου να τεθεί ενισχύ θα χρειαστούν 50 επικυρώσεις και ελπίζω αυτό το όριο να το ξεπεράσουμε του χρόνου. Στην Ευρώπη είμαστε αρκετά προχωρημένοι σε ό,τι αφορά την πολιτική νομοθεσία για τον υδράργυρο, αλλά αρκετοί πολίτες είναι ακόμα ε, εκτεθειμένοι. Οι δέσμοι που έχουμε υποβάλει είναι καταρχάς κανονισμός των συνομοθετών για να ευθυγραμμιστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία με τη σύμβαση και να επικυρώσει η Κομισιόν τη σύμβαση αυτή. Σε ό,τι αφορά την αλληλεία στη Μεσόγειο ε, και τη συνάντηση στην Κατάνια, νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα επιτυχή. Για όσους ε, δεν γνωρίζουν τον υπόβαθρο, ξέρουμε ότι επικρατεί απόλυτο χάος ό,τι αφορά την αλληλεία στη Μεσόγειο. Περίπου 90% των αποθεμάτων ε, τυχάνουν υπεραλίευση. Το πρόβλημα, το κύριο πρόβλημα είναι ότι τη Μεσόγειο τη μοιράζονται κάποια κράτη-μέλη στη Βόρεια Ακτή και άλλες χώρες, ε, τρίτες χώρες, της Βορειοαφρικής στον Νότο. Κάποιε φορέ αυτό χρησιμοποιείται και ω δικαιολογία, γιατί έχουμε κάποια αποθέματα που μόνο κράτη-μέλη αλλιεύουν. Και πάλι παραμένουν ε, αυτά τα προβλήματα με τα αποθέματα. Πρέπει λοιπόν ε, να εξετάσουμε το θέμα της Μεσογείου και από εθνική σκοπιάς και περιφερειακή και ευρωπαϊκής. Τα όσα συζητήσαμε στην Κατάνια ήταν ότι πρώτα πρέπει να εξετάσουμε τα κράτη, μάλλον να συζητήσουμε αυτό το θέμα τα κράτη-μέλη μεταξύ μα. Και εκεί τίθενται τρία ερωτήματα. Πρώτον, αν αναγνωρίζουμε τουλάχιστον ότι υπάρχει πρόβλημα στη Μεσόγειο. Η απάντηση ήταν ναι. Όλοι απάντησαν θετικά. Μετά, Εάν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, θα συμφωνήσουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Και πάλι όλοι απάντησαν θετικά. Και τρίτον, τι θα κάνουμε. Ποια θα είναι τα συγκεκριμένα μέτρα. Προφανώς σταματήσαμε εκεί με το δεύτερο ερώτημα. Γιατί μετά έπρεπε να συμμετάσχουν στη συζήτηση και οι τρίτες χώρες. Έχω προγραμματίσει συνεδριάσεις με την Τουρκία, με την Τινησία, ήδη έχω συναντηθεί με εκπροσώπους της Αλγερίας σε θετικό κλίμα και ελπίζω να συμφωνήσουν και να συμμετάσχουν. Πέραν των χωρών της Μεσογείου, έχουμε και ευρύτερη συνεργασία με την ευρύτερη περιοχή. Η κυρία Μελιόρ μίλησε για την ΕΚΑΠ και την βιοπικιλότητα, εγώ πάντα το θίγω, ανεξάρτητα από το ζήτημα της βιοπικιλότητας, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Ό,τι είναι οι εκθέσεις μας, ε, σε ό,τι αφορά τη φύση, το περιβάλλον, την ενδιάμεση αναθεώρηση, ε, μιλούν για γεωργία και σε σχέση και με το υπέδαφος, ε, την ατμόσφαιρα, το είδωρ και όλους τους τομείς πολιτικής. Εγώ πιστεύω ότι οι γεωργοί θα αποτελέσουν τμήμα της λύσης, γιατί η βιώσιμη καλλιέργεια ωφελεί και τους ίδιους τους γεωργούς. Ήδη πέρσι έχω συναντηθεί με το Γεωργικό Φόρουμ, εκεί μίλησα ανοιχτά. Κάθε γεωργός ε, έχει όφελος ε, να κινηθεί προς ε, μια αλήθιστη πρακτική ως προς τις καλλιεργίες του. Γιατί τελικά θα σημειωθούν και οι ίδιοι από την κλιματική αλλαγή. Εάν λέμε ότι χάνουμε ε, πόρους περιβαλλοντικούς και φυσικούς πόρους, είναι κρίσιμα τα πράγματα. Και εγώ συνομιλώ με τους γεωργούς, όμως θέλω να τους στηρίξω και να συμμετάσχουν και οι ίδιοι σε αυτή τη λύση. Γιατί τελικά είναι προστάτες ε, της βιοπικιλότητάς μας και αν το πράττουν, και εγώ λέω γιατί όχι, να αποζημιωθούν κιόλα. Η κυρία Σχρέιερ και την απώλεια βιοποικιλότητας σε χώροι Natura 2000 για μένα, το έχω πει πολλές φορές, δεν αρκεί μόνο να προσδιορίζεται ένας χώρος ως Natura 2000. Πρέπει να τη χάνει και τις κατάλληλες διαχείρισης. Συχνά μιλούμε για ε, περιοχές Natura 2000 ε, χερσαίες. Όμως έχουμε και αντίστοιχο στόχο και για θαλάσσιες περιοχές Natura 2000. Ενώ Στι χερσαίε περιοχέ Natura 2000 έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλι 4% στι θαλάσσιες περιοχέ. Επομένω, πρέπει ε, να... Ενώ στι χερσαίε περιοχέ μιλούμε μόνο για το πώ θα βελτιώσουμε τη διαχείριση, στη θάλασσα ακόμα παλεύουμε για την ταυτοποίηση αυτών των περιοχών. Συμφωνώ ε, με τα όσα αναφέρθησαν για την επαφή μας με τους Ευρωπαίους πολίτες, ιδίως ότι φορά την πράσινη ανάπτυξη και το καθεξής. Ε, τώρα για τις ε, μονάδες ε, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και το καθεξής, αυτό είναι κάτι το οποίο συζητείται συνεχώς για την Ενεργειακή Ένωση. Κυρίως άλλοι επίτροποι βεβαίως επιλαμβάνουν των θεμάτων, όμως ό,τι αφορά την ενέργεια, από ό,τι ξέρω εγώ πάντα, μάλλον σε ό,τι αφορά εμένα, εγώ πάντα προωθώ ε, τις, βιο... τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί είναι η μοναδική λύση, κατά τη γνώμη μου. Ο μοναδικός τρόπος να προχωρήσουμε. Στις μεταφορές, εντάξει, κάποιοι προσπαθούν να βρουν άλλη λύση με τους, ε, με τους κινητήρες διαφορετική καύσης. Εγώ λέω ξεχάστε όλα αυτά. Πρέπει να στραφούμε προς τις μηδενικέ εκπομπέ. Και, και πάλι, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, εγώ προωθώ κυρίω του ωκεανού. Γιατί όταν μιλούμε για ανανεώσιμες, πάντα αυτά έχουν σχέση με την ηλιακή και την αιωλική ενέργεια. Ενώ ε, στους ωκεανούς μπορούμε να έχουμε και τα ρεύματα και τις ε, τα κύματα. Τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά. Αυτά νομίζω κάποιος μίλησε για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε το μέσο ε, των ερμηνευτικών κατευθυντήριων γραμμών αντί της οδηγίας. Γιατί θεωρούμε ότι είναι ταχύτερο μέσο, ε, μπορούμε να παρουσιάσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές ε, μέχρι τα τέλη του 2016. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη έχει θεσπιστεί μέσω διαφόρων αποφάσεων του δικαστηρίου και ουσιαστικά με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές θα ερμηνεύουμε, θα εξηγούμε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις και θα προωθούμε την εφαρμογή τους και από τα κρατη Σε ό,τι φορά το γλυφοσάτ, είναι το, μια ουσία που χρησιμοποιείται στα ζενιοκτώνα και δόθη έγκριση ε, για την χρήση γλυσοφάτ που λύγει στις 30 Ιουνίου τρέχοντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρω ότι δεν θα με χειροκροτήσετε γι' αυτό, αλλά, ή δεν θα με επικροτήσετε, αλλά ε, η Κομισιόν ανανέωσε αυτή την αδειοδότηση και συνεχίζεται η συζήτηση και με τα κρατημέλη. Ο λόγος είναι ότι η ΕΦΚΑ λαμβάνει, στην αξιολόγησή της λαμβάνει υπόψη και ε, αξιολογήσεις ε, του ΠΟΗ και θεωρεί ότι δεν δικαιολογείται η πλήρης απαγόρευσή του γλυφοσάτ, γιατί υπάρχουν ήδη ε, κριτήρια στην χρήση της ουσίας αυτής, τα οποία είναι ικανοποιητικά. Ε, η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου του αρμόδιου οργανισμού, του ΕΚΑ, θεωρεί ότι πρέπει να ενταχθεί στις μη καρκινογόνες ουσίες. Νομίζω ότι αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι. μπορεί να θέλετε και μια γραπτή απάντηση. Πρόεδρε, για το ψήφισμα ΖΙΚΑ ε, και, τις, ε, και, και τη σχέση... Μάλλον πώ συνδέεται αυτό με τα κουνούπια και τα βαλτόδη ύδατα και ούτε καθεξής. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα και το ίδιο το ψήφισμα. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτά τα ζητήματα, δεν μου απαντήσατε. That's... Yes, probably it's not, my... not under the Νομίζω ότι αυτό δεν υπάγεται στι αρμοδιότητε του κυρίου Επιτρόπου. Είναι ε, ζήτημα δημόσια υγεία. Ναι, αλλά πρόεδρε, τα βαλτόδη ύδατα, καταλαβαίνετε. Ε, και ε, η εκπόνηση του καταλόγου Natura 2000. Γιατί αλλιώς θα έχουμε την κατάσταση που είχαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την μαλάρια. Πρέπει να το εξετάσουμε, αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας. No, I agree with... Συμφωνώ. Δεν λέω ότι δεν είναι δικό μου ζήτημα αρμοδιοτήτων, οπότε δεν με ενδιαφέρει και δεν με απασχολεί. Με απασχολεί και μάλιστα πολύ. Και αν υπάρχει ένα τρόπο να αποτρέψουμε τον ΖΙΚΑ, είναι όπω είπατε κι εσεί, με καλύτερη διαχείριση των υδάτων μα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το προβλέπει και την απασχολεί και μάλιστα για κάθε κράτος μέλος πρέπει να συζητήσουμε λεπτομερώς τις εκθέσεις διαχείρισης των υδάτων. και τα αντίστοιχα σχέδια δράσης για ε, τον πυθμένο των ποταμών, το οποίο ε, αφορά και το ζήτημα που θίξατε. Κάτι το οποίο δεν απάντησα, νομίζω, είναι αυτό που αναφέρθηκε για την Κίνα που απογορεύει την κατανάλωση κρέατος και για την υπευθυνή αλληλεία Νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ, να ευχαριστήσουμε τον Επίτροπο Βέιλα για την παρουσία του εδώ σήμερα και για την ενεργό ε, συνεργασία και βούληση να απαντήσει σε όλες μας τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε και σε ένα λεπτό θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Να δώσουμε ένα λεπτό στον κύριο Πίτροπο να αποχωρήσει για να συνεχίσουμε και εμείς. Έχουμε πολλά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Uh, Ωραία, μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα με το σημείο 5 στην εμισά διάταξη σε ό,τι αφορά τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις για τα όρια εκπομπών, επίσημους ελέγχους, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και την μείωση των εθνικών εκπομπών για τα όρια εκπομπών υπήρξε επίτευξη μιας προσωρινής συμφωνίας με το τελευταίο τριμερή διάλογο στις 6 Απριλίου ε, και καλούμε τους νομοθέτες να δούμε τι είδους ε, δευτερογενής ε, νομοθεσία θα εφαρμοστεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε τα αιτήματα του Συμβουλίου για εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες κινητήρων για τη δυνατότητα αντικατάστασης ορισμένων ε, ε, κατηγοριών κινητήρων. Οδηγηθήκαμε τελικά σε θετικά αποτελέσματα. Προγραμματίζεται ψηφοφορία στις 26 Απριλίου. Για τους επίσημους ελέγχους, ο έκτος τριμερής διάλογος ελευθερών στις 5 Απριλίου ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις για συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα, άρθρων για τον έλεγχο των επίσημων πιστοποιητικών και των εργαστηρίων αναφοράς και υπήρξαν συγκεκριμένες διευκρινήσεις. Σε επικοδομητικό κλίμα έγιναν οι συζητήσεις και υπήρξε συμβαστική λύση για περισσότερα πολιτικά ζητήματα. Ο 7ος ε, τριμήρης διάλογος θα λάβει χώρα αύριο για τα ιατροτεχνολογικά και τα IVF, τα in vitro τεχνολογικά προϊόντα. 7 Απριλίου έκλεισαν πολλά σημαντικά ζητήματα και έτσι τα μέρη θεωρείται ότι έχουν σημαίνει σημαντική ε, πρόοδο. Η πρόταση ε, της Κορεπέρ στις 21 Μαρτίου έκλεισε συμφωνία για συγκεκριμένα εργαλεία και σε ό,τι αφορά τον κανόνα 6, Και η Κομισιόν έκανε ορισμένε προτάσεις ε, για ε, συγκεκριμένους εργαστηριακούς ελέγχους in vitro και τα δύο θα πρέπει να τα εξετάσει Κοινοβούλιο και Συμβούλιο και να ξαναμπούν στο, στη μεσοδιάταξη για ένα το τριμερή διάλογο. Εκκρεμούν ορισμένα ζητήματα στα in vitro κάποια στοιχεία του κεφαλαίου 6, κανόνες ε, συνταγογράφησης, ταξινόμησης 1, 4 και 5, το new Patient Testing, μετά έχουμε τον επόμενο τεμερή διάλογο στις 11 ε, Μαρτίου. Για την οδηγία ΝΕΚ, e ο δεύτερος τεμερής διάλογος έλαβε χώρα στις ε, 5 Απριλίου υπήρξε πρόοδος ό,τι αφορά τη συμφωνία για λιγότερο φιλογόμενα ζητήματα. Ε, για την καθαρή ατμόσφαιρα και να υπάρξει αντίστοιχο ταμείο και φόρουμ. Ε, εξετάστηκαν διάφορα ζητήματα συμπεριλαμβανομένου του παρατήματος 2. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στα επόμενα σημεία της διάταξης έκθεση τη Επιτροπή προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία το 2014. Ο κύριος Στέβεναντ είναι εδώ μαζί μας από την αρμόδια μονάδα στη Γενική Διεύθυνση ε, Υγείας και Καταναλωτών. Να του δώσουμε το λόγο για να μας παρουσιάσει την έκθεση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι μιλούμε για την έκθεση που δημοσιεύει κάθε χρόνο η Κομισιόν σχετικά με τις ε, δράσεις ε, των αρχών ελέγχου για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ε, που προβαίνουν σε ιονίζουσα ακτινοβολία επί συγκεκριμένων προϊόντων και για τους ελέγχους που επιβάλλονται στα αυτά τα προϊόντα μετά τη θέση εμπορία. Η Κομισιόν θυμίζει λοιπόν τον κατάλογο των κρατών μελών που έχουν τέτοιε εγκαταστάσει, 13 είναι αυτά Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Εστονία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, κάτω Πολωνία, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον και η Νορβηγία έχει μια τέτοια εγκατάσταση. Ο συνολικός όγκος στην Ιερακή Ένωση το 2014 ήταν 5.500 τόνοι. Λιγότερο από τις προηγούμενες ε, χρονιές, 20% μείωση το 2013. Η επεξεργασία αυτή, θυμίζω, αποβλέπει στην, ε, καταστροφή κάποιων παρασίτων ή μικροβίων, ε, κυρίως τα στους καρπούς. Το κείμενο έχει επιτρέψει την εναρμόνιση μόνο συγκεκριμένων είδων, προϊόντων, βότανα, λαχανικά, εποχής, αλλά ξηρά, σε ξηρά μορφή και όχι σε νοπή. Και έχουμε εθνικές εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις για συγκεκριμένα προϊόντα στο Βέλγιο, στην Τσεχία, την Γαλλία, την Ιταλία, την κάτω, τις κάτω χώρες, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ των προϊόντων αυτών, εθνικής φύσεως, είναι λαχανικά, φρούτα, αλλά και κρέας. Όπως και βατραχοπόδαρα. σχετικά με τα προϊόντα που έχουν ε, δεχθεί τέτοια ακτινοβολία, στην ουσία στην Ευρώπη μιλούμε για τα παντραχοπόδαρα. Είναι το 55% του συνόλου. Σε όγκο. Το δεύτερο με 16% είναι τα σφάγια πουλερικών. Και το τρίτο είναι τα χόρτα βοτανικά. Τα βότανα, με συγχωρείτε, και τα, χορτα... τα βότανα τα αρωματικά χόρτα. Το Βέλγιο και η Ολλανδία είναι το 85% της επεξεργασίας, με το Βέλγιο 60% και 24% η Ολλανδία. Σχεδόν. Το τρίτο πολύ μακριά με 8% είναι η Γαλλία. Κατά το του 2014 έγιναν 6.000 περίπου δοκιμές έλεγχη στα κράτη-μέλη με 98% θετικά αποτελέσματα, 1% αρνητικά και 1% ασαφή λόγω των μεθόδων που ακολουθήθηκαν. Τα τεστ αυτά έγιναν στα προϊόντα που είχαν τεθεί σε εμπορία. Τα αρνητικά αποτελέσματα μπορούσαν να οφείλονται είτε στην επισήμανση, γιατί και το θεσία ήταν ασαφής, είτε στο γεγονό είτε στο γεγονός ότι ο έλεγχος δεν έλαβε χώρα σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, αλλά οδήγησε στην απόσυρση από την αγορά, εκτός από τις περιπτώσεις ετικετοθεσίας όπου ο παρασκευαστής μπορούσε να ε, επιλέξει την ε, νέα επισήμανση και τη νέα θέση εμπορία. Τώρα η κατανομή των ελέγχων είναι σημαντική. Η Γερμανία έχει δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε εξακριβώσει και τους ελέγχους αυτούς και σχεδόν στο ίμιση των προϊόντων που, των προϊόντων που δοκιμάστηκαν η έλεγχη αυτή έγινε στην Γερμανία. Επίσης η Ιταλία και η Ολλανδία δίνουν μεγάλη σημασία στο ελέγχους αυτούς γιατί μεταξύ τους μοιράζονται το 70% των ελέγχων που έγιναν το 2014. Ιδού το περιεχόμενο της εκθέσεως αυτής και ίσως ε, θα δώσω τώρα το λόγο στα μέλη και είμαι στη διαθεσή σας για απαντήσεις. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στους συναδέρφους, εάν κάποιος θέλει να θέσει ε, κάποια ερώτηση, έχει τη δυνατότητα. Κύριο Χόισλινγκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Το θέμα αυτό δεν συζητείται πολύ, είναι όμως ενδιαφέρον όσον αφορά την η οντίζουσα ακτινοβολία. Υπάρχει ευρύ φάσμα δόσεων ακτινοβολίας. Είναι δύσκολο να ενημερωθεί κανείς σωστά σχετικά με τις δόσεις διάφορα κράτη-μέλη. Έχουν, ε, δώσει, ε, έχουν αιτιολογήσει ε, τη, την έλλειψη ελέγχων με τρόπο κάπως περίεργο, ότι δεν είχαν αρκετό ανθρωπίνα δυναμικό και τέτοια. Και επίσης ε, στην έκθεση δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές. Έχω και μια συγκεκριμένη ερώτηση που έχει να κάνει με τη σχέση ανάμεσα στην ε, ιοντίζουσα ακτινοβολία και την ε, μικροβιακή αντοχή. Μπορεί δηλαδή η οντίζουσα ακτινοβολία να οδηγήσει σε ανθεκτικά μικρόβια. Και επίσης τι έλεγχος γίνεται όσον αφορά την ιοντίουσα ακτινοβολία στα τρόφιμα. Ε, η έκθεση δεν συμπεριλαμβάνει συμπεράσματα. Τι δηλαδή θα πρέπει να κάνει η Κομισιόν για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχουμε δεδομένα εισαγωγών και εξαγωγών, διότι δεν είναι μεταξύ των στοιχείων που υποτίθεται ότι λαμβάνει η Κομισιόν από τα κράτη. για την μικροβιακή αντοχή. Για να είμαι ειλικρινής δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η την ακτινοβολία καταστρέφει τα μικρόβια. Αλλά επιστημονικός πώς, κατά πόσον θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο ή επιρροή επί της μικροβιακής αντοχής έχω κάποιες αμφιβολίες, θα πω απλώς, αλλά θα θέσω το ερώτημα σε αρμοδιότερους. Για το bird's eye view, η Κομισιόν ε, καταθέτει μια έκθεση κάθε χρόνο, μια έκθεση που επικεντρώνεται βεβαίως στα μεγέθη και τους αριθμούς, αλλά θα προσπαθήσουμε να εξεγάγουμε κάποια συμπεράσματα και να δούμε σε ποιο μέτρο θα μπορούσαμε να ξαναδούμε αυτήν την, ε, το πλαίσιο νομοθεσίας που ναι έχει τα χρονάκια του. Αλλά θα έχουμε τα αποτέλεσματα πρώτα του, των αρχών του 2015 για να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Αν ε, δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο και να περάσουμε στο επόμενο. Δεν έχει φτάσει ακόμα όμως εκπρόσωπος της Κομισιόν για αυτό το θέμα. Ας κάνουμε μια λιγόλεπτη διακοπή περιμένοντας ε, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα κλείσουμε εδώ τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ξεκινήσουμε αύριο το πρωί, ως συνήθως, στις 10.30 μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών. Σας ευχαριστώ πολύ, θα το πούμε αύριο.